Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αν συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαι σίγουρος πως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα έρθουν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που θα γίνουν. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους και θα ήθελα να καλωσορίσω και τα μέλη του πάνελ. Βεβαίως θέλω να καλωσορίσω ε, και τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Ανάπτυξης, όπως επίσης και τον Αντιπρόεδρο ε, της Επιτροπής αυτής. Το πρώτο πάνελ έχει να κάνει με τα διδάγματα που αποκτήσαμε από την έκτη παγκόσμια αξιολόγηση της ε, ε, αναπτυξιακής βοήθειας σε ε, αντάλλαγμα για εμπορικά πλονεκτήματα, το Aid for Trade, και την αξιολόγηση που έγινε στην ε, Γενέβη πρόσφατα. Έχω τον κύριο Ρούμπιχ κοντά μας σήμερα, ο οποίος είναι συνάδελφος και ο οποίος ήταν ε, παρόν στην ε, συνδιάσκεψη αυτή. Θα συζητήσουμε και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα και θα δούμε τι σημαίνουν για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στο χώρο αυτό. Ξέρετε πως η πρωτοβουλία Aid for Trade ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2005 ε, στο Hong στην Υπουργική συνδιάσκεψη εκεί και αποτελεί ένα συμπληρωματικό στοιχείο στο θεματολόγιο της Ντόχα. 300 δις περίπου ε, δολάρια έχουν εκταμιευθεί ε, για το θέμα αυτό και είναι 146 οι αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες έχουν βοηθηθεί μέσω αυτής της διευκόλυνσης στην Αφρική και στην Ασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην εχμή των όσων προσφέρουν τέτοιου είδους αναπτυξιακή βοήθεια με 12,7 δις το 2014 δηλαδή το 30% περίπου της συνολικής ε, βοήθειας που προσφέρεται. Τώρα όμως χρειάζεται εμείς να εξελίξουμε το πλαίσιο υπό το οποίο προσφέρεται η βοήθεια αυτή και θα πρέπει ε, να έχουμε την προσπελασιμότητα και τη βιωσιμότητα, όπως επίσης το γεγονός πως είναι ανοιχτή σε όλους αυτή η βοήθεια ως βασικές αρχές που θα διέχουν το πλαίσιο. Νομίζω πως ε, το μόνο που χρειάζομαι είναι να συνδέσω τη σημερινή ε, ακρόαση με την ε, συνάντηση της Ινταχτές που μιλήσαμε για την Αφρική και η Ευρωπαϊκή Επίτροπη χτες μας είπε ότι τα επόμενα 20 χρόνια χρειαζόμαστε 18 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για να κατέτος ε, για να ξεπεράσει η Ήπειρος αυτή τα προβλήματά της και σήμερα δεν βρίσκονται στοιχώς στα 18 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης κατέτος αλλά στα τρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το θέμα και είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το μεταναστευτικό και θα το κλείσω εκεί δίνοντας το λόγο ε, στον συνάδελφο που είναι αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης για να ε, συνεχίσει ε, ε, μετά τα όσα σας είπα και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ στα γρήγορα να σχολιάσω τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος της ΙΝΤΑ. Να σας πω πως σε κάποιες χώρες οι σχέσεις μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης έχουν γίνει απόλυτα κατανοητές. Εγώ είμαι Φιλανδός και για πολύ καιρό Ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό χαρτοφυλακίων ε, στην κυβέρνησή μας και είναι πάντα ο Υπουργό που για θέματα εμπορίου που έχει και τα θέματα ανάπτυξης στο ίδιο χαρτοφυλάκιο. Να σας πω πως τη μερίδα του Λέοντος στα ανεπτυξιακά κονδύλια την κατευθύνουμε στην στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών έτσι ώστε να ε, ενισχυθούν οι εμπορικέ του δυνατότητες οπότε ε, το να περάσουμε μετά στη σύνδεση Aid for Trade δεν είναι μόνο ένα στρατηγικό στόχος αλλά είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι και σε οικονομικό επίπεδο ε, είναι απαραίτητο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας οι, αναπτυξιακοί. Είναι πάντα και πρωταρχικά η καταπολέμηση της ένδυας. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να ξεπεράσουν τη φτώχεια ε, που τους μαστίζει. Θα πρέπει ε, στρατηγική μας λοιπόν να συνδυάζεται με τη συνολική πολιτική σχετικά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να ακούσω από τα μέλη του πάνελ τα διδάγματα τα οποία έχουμε αποκτήσει, τις ευκαιρίες αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Σας δίνω λοιπόν και πάλι ε, το μικρόφωνο αγαπητέ συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Όπως συμφωνήσαμε, ε, τη στιγμή που προετοιμάζαμε τη σημερινή συνάντηση και πριν δώσουμε το λόγο στα μέλη του πάνελ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λούμπιχ, ο οποίος, Ρούμπιχ, με ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την διάσκεψη που έγινε στη Γενέβη, στην έκτη διάσκεψη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή ακριβώς είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον των συμπολιτών μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, και να δούμε πώς μπορούμε με την ε, αναπτυξιακή βοήθεια να στηρίξουμε. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να έχει κατανάλωση, θα πρέπει να στηρίξει την παραγωγή. Είναι τα καταναλωτικά δικαιώματα τα οποία είναι σημαντικά και θα πρέπει να επιλέξουμε ε, τα προϊόντα τα οποία θεωρούμε ότι είναι τα καταλληλότερα για μα Είναι σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη και στι εισαγωγές και στι εξαγωγέ, γιατί αν μπορεί κανείς καλύτερη ποιότητα και πιο φθηνή ε, να, και πιο φθηνά να αποκτήσει ε, ένα αγαθό από κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, τι κάνεις, αποκτάς μεγαλύτερη αγοραστική αξία, ε, δύναμη και βεβαίως το ίδιο ισχύει και αν κάνεις εξαγωγές, γιατί πληρώνεσαι ένα μισθό, ο οποίος ε, αυξάνεται με την αύξηση των εξαγωγών, άρα και εκεί η αγοραστική σου δυνατότητα αυξάνεται. Άρα λοιπόν όταν προχωράς και σε εισαγωγές και σε εξαγωγές, τότε είναι διπλό το πλεονέκτημα για τους καταναλωτές. Άρα λοιπόν θέλουμε να προκρίνουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, όχι μόνο των μεγάλων βιομηχανιών και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το πλεονέκτημα που θα προσφέρει το εμπόριο για όλους τους πολίτες και τους δικούς μας και των υπολείπων χωρών. Ξέρετε πως στην, ε, στη διάσκεψη του Σιάτελ, εκεί που ξεκίνησε το θέμα αυτό, ε, τα πράγματα ήταν κάπως περίπλοκα. Κανείς δεν ήταν ακριβώς έτοιμος να διαπραγματευτεί τα θέματα αυτά. Αλλά ο ΠΟΕ μας έχει δείξει πως είναι πιθανό και είναι δυνατόν να κάνει κανείς να σημειώσει κανείς πρόοδο. Ε, πήγαμε στο Χονγκ Κονγκ και εκεί αποκτήσαμε το θεματολόγιο για το εμπόριο, για, τα, για τις τρεις πυλώνες, διευκόλυνση εμπορίου, aid for trade και ε, για τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες. Το θέμα αυτό είναι και το πιο σημαντικό, δηλαδή εμπορικά ανταλλάγματα ε, μέσω ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι πολλές οι χώρες που έχουν λάβει αυτή ε, τη βοήθεια. Το 41% πήγε στην Ασία, στην Αφρική ε, πήγε το 38% αυτής της βοήθειας και αν έχετε δει και τα στοιχεία από χθε, θα διαπιστώσετε πως έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το Ταμείο για την Αφρική Κάτι το οποίο στήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είπαμε πως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Αφρική και το Aid for Trade είναι πολύ σημαντικό σχετικά. Και το 27% του ε, συνολικού προπολογισμού πάει στις λιγότερο αναπτυγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουμε πως οι εκταμιεύσεις έχουν πάει σε κυρίως τέσσερις ε, ε, κλάδους στην, ε, στις μεταφορές και στην αποθήκευση, στην παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας είναι η βάση κάθε πλούτου, γιατί παραγωγή ενέργειας, παραγωγή νερού κτλ. Και μετά έχουμε και τη γεωργία, όπου έχουμε το ελάχιστο που θα πάει μετά τη γεωργία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στην ε, στον τραπεζικό κλάδο και εδώ θέλω να τονίσω τη σημασία που αποκτούν καθημερινά περισσότερο το internet banking και οι άλλες σχετικές υπηρεσίες από το διαδίκτυο. Είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός. Είπαμε ότι έχουμε φτάσει περίπου τα 27 δις από το 2014 και μετά και στη διάσκεψη αυτή κάναμε και μια προσπάθεια παρακολούθησης που πήγε πολύ καλά και από τις δύο πλευράς, δηλαδή και αυτοί οι οποίοι έλαβαν τα κονδύλια και αυτοί οι οποίοι ε, τα προσφέρουν και είναι ένα είδο αυτοαξιολόγηση. Έχουμε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε πώς μπορούν οι προσπάθειες ε, συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού κλάδου να φέρουν αποτελέσματα και να έχουμε επιτυχή project τα οποία ε, μετά θα αναλυθούν. Αυτά τα βρήκαμε στην έκθεση ε, που παρουσίασε η διάσκεψη όταν τελείωσε και νομίζω ότι είναι μια έκθεση που πρέπει να τη διαβάσουμε. Έδειξε σε πολιτικό επίπεδο ποιε είναι οι πραγματικέ επιτυχημένε ε, περιπτώσει και έχουμε και τα infographics που κάνουν μια απογραφή των διάφορων δραστηριοτήτων, το πώ αυτέ εξελίχθηκαν. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Και νομίζω πως και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα εργαλείο που θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στις περαιτέρω συζητήσεις που θα κάνουμε. Θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια καλύτερη στόχευση και στην Αργεντινή θα δούμε πώς μπορούμε εκεί να βελτιώσουμε ε, τα όσα προσπαθούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί και με ε, την ε, Διεθνή Ένωση Κοινοβουλευτικών που έχουμε ιδρύσει με τη συνάδελφο και που συναντιόμαστε μία φορά τουλάχιστον το χρόνο όταν γίνονται οι διπολικές συναντήσεις με, φιλ, με συναδέλφους βουλευτές από όλο τον κόσμο. Την τελευταία φορά ήμασταν 400 βουλευτές με τους ε, υπουργού Εμπορίου και η Steering ε, Επιτροπή, η Επιτροπή ε, του ΠΟΕ είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και τα θέματα αυτά τα συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια πολυμερή διάσταση και για το θέμα αυτό νομίζω ότι για τι πολυμερεί, αλλά και για τι διμερείς ε, συμφωνίε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με τη χειραφέτηση των, γεγονο... γυναικών, με τη ευκόλυνση του εμπορίου, με την ψηφιακή ατζέντα και επαναλαμβάνω στη Γενέβη οι συμμετέχοντες ήταν γύρω στους 1500 και αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά. Πάνω από 50 διαφορετικές εκδηλώσεις, μια πολύ, ένα πολύ ε, μεγάλο πεδίο εφαρμογής, έτσι ώστε οι λιγότερο αναπτυγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να βρεθούν τελικά σε μια καλύτερη κατάσταση. Τα κομβικά σημεία ε, στα οποία συγκεντρώσαμε τις προσπάθειές μας είναι ο τρόπος που θα μας επιτρέψει να, να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάος χάσμα, με συγχωρείτε, τη χειροθέτηση των γυναικών. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα κατά τη γνώμη μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πολύ δραστήριοι σε, αυτό το, σε αυτή την εργαλειοθήκη ε, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να χειραφετήσουμε τις γυναίκες ως σημείο κλειδί για να βελτιωθεί η κατάσταση των χωρών αυτών. Και για πρώτη φορά Μιλήσαμε και για την ε, εφαρμογή της Συμφωνίας Διευκόλυνση του Εμπορίου. 22 Φεβρουαρίου 2017 έγινε η σχετική συνάντηση και εκεί αντιμετωπίσαμε μία περίπτωση που πέρασε από τον ΠΟΕ είναι τα σύνορα μεταξύ Κένιας και Ουγκάντα και τι έκανε σε πρακτικό επίπεδο επιτόπου η, η Συμφωνία για την Εμπορική Διευκόλυνση. 210 φορτηγά περνάνε καθημερινά αυτό το σημείο στα σύνορα ε, έκτοτε, κάτι το οποίο λοιπόν ε, πόσο καλό ήταν το ότι ο χρόνος διέλευση των συνόρων για τα φορτηγά αυτά μειώθηκε κατά 79%. Είδατε πόσο σημαντικό είναι. Και ήρθε και ο αναπληρωτής ε, Πρωθυπουργό τη Γκάμπια, όπω επίση και ο Υπουργό Εμπορίου. Είναι μια καινούργια κυβέρνηση και με χαρά του υποδεχτήκαμε. Είναι μια νέα διάσταση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να βλέπουμε πω αυτή η συνδιάσκεψη αξιολόγηση για πρώτη φορά μας συμπεριλαμβάνει και γι' αυτό ευχαριστώ τον ΠΟΕ και πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή θα είναι πολύ ε, κερδοφόρος και για το μέλλον. Σε ευχαριστούμε Πάουλ για όλες αυτές τις πληροφορίες και τα νέα στοιχεία και τώρα να ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ αυτής της ακρόασης. Στην ακρόαση αυτή λοιπόν θέλω να καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Μάικλ Ρόμπερτ, ο οποίο είναι διευθυντή του Aid for Trade τη Υπηρεσία για την Ανάπτυξη στον ΠΟΕ. Θέση την οποία κατέχει από το 2009. Στην έκτη παγκόσμια αναθεώρηση του Aid for Trade συμμετείχε πλήρω βέβαια. Από το 2001 έχει ξεκινήσει συνεργάζεται στο θέμα αυτό, όταν ε, δούλευε στην ε, υπηρεσία για τα αγροτικά και τα τρόφιμα στον ΠΟΕ. Έχετε το λόγο για 7 με 8 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, συμπρόεδρε. Βλέπω ότι το PowerPoint λειτουργεί ήδη. Όπως είπατε στις προκαταρκτικές σας η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, αποδίδουν το 1 τρίτο της συνολικής βοήθειας για το εμπόριο σε σχέση με άλλους πολυμερείς οργανισμούς ε, και άλλες φορείς είναι μεγάλο το μερίδιο. Η στατηγική η γη του Aid for Trade δείχνει τις νέες ανησυχίες για την ανάπτυξη και τη στρατηγική μας και σε αυτό το τοπίο είναι η καταλληλότερη στιγμή για να σας ενημερώνω για τα πορίσματα της 27ης αναθεώρησης. Όπως είπε και ο συνάδελφός σας ο κύριος Ρούμπιχ, με κάποια στατιστικά στοιχεία για την παγκόσμια αναθεώρηση. Τα βλέπετε στη διαφάνεια, βλέπετε κάποιους αριθμούς από αυτούς που αναφέρατε. Στον λιγοστό χρόνο που έχω, θέλω να σταθώ σε τέσσερα βασικά θέματα. Θέματα τα οποία και εσείς εντοπίσατε, την ψηφιακή διασύνδεση, την χρηματοδότηση, τη διευκόλυνση για το εμπόριο και την ανάληψη ευθύνη. Θα προσπαθήσω να τα αναπτύξω. Ευχαριστώ όμω πολύ για τα θερμά λόγια καλώ ορίσματο για την έκθεση αυτή και να πω ότι τρεις από τους συντάκτες της έκθεση που κάθονται δίπλα μου ο ένας και οι άλλοι που θα έρθει στη διάσκεψη μαζί μας έχουν εργαστεί εντατικά για το θέμα αυτό, για την ψηφιακή διασύνδεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κοιτάζει την νομοθετική ε, αρχιτεκτονική της νέας ψηφιακής αγοράς σε διαφορετικά στάδια. Για την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο οργανισμός ITU, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τις Τηλεπικοινωνίες, ε, μας λέει ότι υπάρχουν 3,8 δις άνθρωποι εκτός ίντερνετ ε, και ιδίως στην Αφρική. Υπάρχει ψηφιακό χάσμα, αλλά υπάρχει και θέμα πρόσβαση στην αγορά. Όσοι δεν είναι ε, online, δεν έχουν επικοινωνική πρόσβαση, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται ε, παγκοσμίω στην ηλεκτρονική αγορά. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο σίγουρα θα το αναπτύξει περαιτέρω η κάτι στα σχολεία του. Είναι βεβαίω ε, τροχοπέδι αυτό στην οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο και βεβαίω ιδίω για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Υπάρχουν θετικέ εμπορικέ ενέργειε που μπορούν να αναλάβουν οι αναπτυσσόμενε χώρε για να επηρεάσουν την προσφορά και ζήτηση στην όλη ε, ισορροπία. Πρώτα απ' όλα η διαθεσιμότητα της ψηφιακής διασύνδεσης και το κατά πόσον είναι χαμηλές τιμές. Αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα στα σχόλια. Η ιδέα ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση της ζήτησης έχει να κάνει με το ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες η Παγκόσμια Τράπεζα καλύπτει μόνο το 50% ε, ε, του πληθυσμού, αλλά οι υπόλοιποι μόνο μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Εδώ βλέπετε κάποια οικία σας πρόσωπα. Η Παγκόσμια Σύνοδος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, για να πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είναι μια διαδικασία που οδήγησε στην εκπόνηση εθνικών προγραμμάτων για την διασύνδεση στα συστήματα επικοινωνία και πληροφορία για τι ανεπτυσσόμενε χώρε, όμω απαιτείται χρηματοδότηση για αυτά. Η έρευνα που έκανε όσα για την παγκόσμια αναθεώρηση του Aid for Trade δείχνει ότι χρειάζονται 536 εκατομμύρια δολάρια του Aid for Trade. Αυτά πήγαν για τη διασύνδεση ICT το 2016 μεγαλύτερη χρηματοδότηση στον κλάδο αυτό προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα από τα συμπεράσματα λοιπόν προέρχονται από την ε, διάσκεψη είναι να δούμε κατά πόσον αυτή η βοήθεια σε ευρώ, σε δολάρια μπορεί να είναι καταλήτης για επενδύσεις ε, ε, επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και αυτό μας φέρνει πίσω στις δηλώσεις του Επιτρόπου Μιμίτσα για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και θα πρέπει να τα δείτε και εσεί στι επιτροπέ σα για την αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Aid for Trade. Αλλά στον όσα σκεφτόμαστε το όλο θέμα βλέποντα τι προτάσει που έχουν γίνει σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την διευκόλυνση των επενδύσεων ε, εντό του ΠΟΕ. Ο κ. Ρούμπιχ ανέφερε το τι έγινε με, το, με την διέλευση Μπούζια Μπόζακ ε, στην Αφρική αυτή είναι τη συγκεκριμένη περίπτωση και παράδειγμα, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά σε σχέση με παρόμοιε περιπτώσει. Ένα από τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε με την παγκόσμια αναθεώρηση είναι το πώ η διευκόλυνση για το εμπόριο μπορεί να διασυνδέσει τα θέματα αυτά με το ηλεκτρονικό εμπόριο Εάν σκεφτείτε το ηλεκτρονικό εμπόριο, μιλάμε για ταχυδρομικά πακέτα περισσότερο παρά για μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια, σε κοντέινερ. Είναι διαφορετική λοιπόν η σκέψη για τους δασμούς και το πώς μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μια υποσημείωση που ίσως σας ενδιαφέρει, που θα μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια ενδεχομένω, είναι ότι κάποιες από τις συζητήσεις είχαν να κάνουν με τη διευκόλυνση για το εμπόριο και τις σχετικές βελτιώσεις που μπορούν να ε, συμβάλλουν ακόμη και στην ανακούφιση από φυσικές καταστροφές. Το τέταρτο θέμα είναι η ανάληψη ευθύνης. Η ενίσχυση. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διάσκεψη είναι ότι χρειάζεται περισσότερο από ψηφιακή απλώ διασύνδεση για να υπάρξει συμμετοχή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. υπάρξουν δεξιότητε, χρηματοδότηση, το κατάλληλο περιβάλλον και όλα αυτά είναι εχθρικά όμως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε σίγουρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τις γυναίκες και όσες επιχειρήσεις έχουν ε, γυναίκες σε διευθυντική θέση. Θα πρέπει λοιπόν οι φορείς και οι κυβερνήσεις να λάβουν υπόψη και τη διάσταση του φύλου στο πρόγραμμα Aid for Trade και πώς προχωρούμε, πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα στοιχεία και ερευνές και αποτελέσματα για το θέμα αυτό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα λοιπόν ε, στην αναθεώρηση του Aid for Trade και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποφασίσει να επικαιροποιήσει τη στρατηγική του Aid for Trade και για σκοπούς χρηματοδότησης και για το πόσο βαρύνει η φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΠΟΕ. Είναι οικίε οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το ξέρετε, έχουν αναφερθεί. Έχουμε και έναν οδικό χάρτη με ε, όριο το 2030. Και με αυτά τα σχόλια επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην ενεθρώση της στρατηγικής σας Aid for Trade και ελπίζω να τα πάτε καλά σε αυτό το σημαντικό θέμα. Uh, thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ε, παρατηρήσεις που κάνατε σε ό,τι αφορά το συντάκτη της αναθεώρησης. Ε, και τώρα να περάσουμε στον δεύτερο ομιλητή, ο κύριος Λάμερσεν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ε, στον ΩΣΑ από το 97 στην Διεύθυνση Ανάπτυξης που συνδράμει και βοηθά την Σχετική Επιτροπή και είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων για τα συνδέματα αυτά μαζί με τον κύριο Ρόμπερτς ήταν υπεύθυνο για τη δημοσίευση του κειμένου στη Γενέβη 2. Του δίνω λοιπόν το λόγο περίπου για την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι η πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στην Κίνα της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ανάπτυξη του οικολογικού αποτυπώματος και θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε την ίδια γλώσσα, θα πρέπει να συνεννοούμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για το παρελθόν, για το μέλλον και ενδεχομένω το τι μας επιφυλάσσει, μάλλον το παρελθόν, το παρόν και το τι μας επιφυλάσσει και το μέλλον σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της ε, συνεδρίας της αυτής. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Aid for Trade είναι ότι περιλαμβάνει ε, μια παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των πρωτευουσών σε μια κοινή ατζέντα. Βάσει της διαφάνεια, και της λογοδοσίας μπορεί να υπάρξει διάλογος προκειμένου να βοηθήσουμε πραγματικά τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν ε, το δυναμικό τους. Με εμπορικές συμφωνίες, για παράδειγμα, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο όφελος Τη Παγκόσμια Πρωτοβουλία Aid for Trade είναι μια πολύ ευέλικτη ατζέντα η οποία εναρμονίζεται πάρα πολύ με τα, τους στόχους της του εμπορίου. Το 2009 μετά την οικονομική κρίση το επίκεντρο ήταν να δούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε το 2011. Θέλαμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιτεύγματα. Στη συνέχεια θελήσαμε να υπάρξει ένας σύνδεσμος ε, μια σύνδεση μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών και των ε, αναπτυγμένων χωρών. Γιατί θέλαμε λοιπόν να δώσουμε μια ευκαιρία βιομηχανοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ύστερα αντιληφθήκαμε ότι αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι να μειώσουμε το εμπορικό κόστος που είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτο και υψηλό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις αγεργικές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Και ε, ουσιαστικά δεν αναπτύσσονται όσο θα θέλαμε στις χώρες όσα. Και τέλος, το είπαν και οι συνάδελφοι, θα το αναφέρουν και άλλα, άλλοι συνάδελφοι στο μέλλον, είναι το θέμα της συνδεσιμότητας σε ό,τι αφορά απομονωμένες περιοχές. Ήταν πολύ αποτελεσματική η πρωτοβουλία, θεωρώ. Το εμπόριο πλέον ε, δεν είναι, στο εμπόριο δεν πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην κατάρτιση προγραμμάτων και στρατηγικών σχεδιασμών και υπάρχει εναρμόνιση βάσει της προτεραιότητας αυτής. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, το ανέφερε και ο συνάδελφος, ε, ο συνάδελφος ο κ. Ρούμπιχ, οι ροές του Aid for Trade προς τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες έχουν φτάσει από 23 δις σε 53 δις πλέον. Είναι σημαντική υπερδιπλασιασμός η αύξηση αυτή των ε, πόρων. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο τα χρήματα και οι πόροι, αλλά και το κατά πόσο πετυχαίνουμε τα αποτελέσματα. Και πολλές ακαδημαϊκές ε, μελέτες καταδεικνύουν ότι και μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από τις εκάστοτε χώρες, αλλά γίνονται σχετικές αναλύσεις. Όλες καταδεικνύουν ότι ένα δολάριο στο Aid for Trade δημιουργεί 8 δολάρια στις υπόλοιπες χώρες και 20 ε, δολάρια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί από αξιολογήσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, όλες πολύ θετικέ. Και από μελέτες περιπτώσεων που καταδεικνύουν ότι πραγματικά το Aid for Trade επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων τόπου Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι χρειάζεται καλύτερο aid for trade από ζητείται από τη σχετική ατζέντα. Δεν θέλουμε μόνο μεγαλύτερο όγκο, αλλά και καλύτερο aid for trade από το που είπε ο συνάδελφο πριν από λίγο. Ότι αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται σε μία νύχτα Κοιτάξτε για παράδειγμα τη διευκόλυνση, τη εμπορικέ διευκόλυνση. Ε, καλό παράδειγμα, αλλά χρειάζεται διαλειτουργικότητα, περιφερειακή συνεργασία, υποδομέ. Αυτά παίρνουν χρόνο. Και κοιτώντα λοιπόν παραδείγματα όπω το Βιετνάμ, το Παγκλατέ, Ουγκάντα, Κάνα, όλα αυτά έγιναν και επιτεύχθηκαν μέσα σε 10-15 χρόνια. Θα πρέπει τώρα να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το τι συμβαίνει. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αξιολογούμε προγράμματα όπου υπάρχει σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν διάφορε τέτοιε περιπτώσει, ε, Αυτά τα PPPs δουλεύουν. Πρόκειται πραγματικά για εμπορικού τομεί ε, τομεί βιομηχανοποίηση όπου θέλει ο ιδιωτικό κλάδο να συνεργαστεί με το δημόσιο. Πώ δημιουργούμε λοιπόν τέτοια περιφερειακά αποτελεσματικά προγράμματα αν βασίσουμε τις στρατηγικές μας, τις εθνικές προτεραιότητες, πώς λαμβάνουμε υπόψη και τις περιφερειακές προτεραιότητες και πώς ως δωρητής μπορεί κανείς να εναρμονίσει τις ανάγκες του. Ο Μάικλ μίλησε για τη χρηματοδότηση. Πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία, ήταν επιδοτήσεις 64% ε, το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. 60% είναι δάνεια και 4% μόνο είναι επιδοτήσεις. Αυτό είναι το θυμόμαστε, 60% των LDCs δεν έχουν πλέον άλλο οικονομικό χώρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Μιλάμε και για γεωργικές δραστηριότητες, για να δημιουργηθεί στον ιδιωτικό κλάδο κέρδος, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε τι γίνεται και να μην υπάρξει στρέβλωση της ενιαίας αγοράς. Ε, δεν έχω και πολύ χρόνο θα περάσω στο επόμενο θέμα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι δεσμεύσει και του περιορισμούς του διάφορου τομεί. Κοιτάμε ποιο είναι και η σύνδεση μεταξύ εμπορίου και επενδύσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ατζέντα αυτή ε, θα είναι μακροπρόθεσμη. Θέλει όραμα, θέλει επένδυση, υπομονή και επιμονή. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα επιτέχματα πολύ σημαντικά τα οποία έχουμε ήδη πετύχει. Γιατί μια αναπτυσσόμενη κοινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι εμείς χτίσαμε αυτή τη γέφυρα. Πιο σημαντικά είναι νοσοκομεία, σχολεία. Αλλά μακροπρόθεσμα είναι δύσκολο να γίνει αυτή η σύγκριση. Ποιο πρόγραμμα είναι πιο ωφέλιμο, ποιο έργο είναι πιο ωφέλιμο. Για το μέλλον λοιπόν υπάρχουν τα έργα τα οποία ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και ο Μάικλ το ενδιαφέρει ότι βασικά ο πρώτος στόχος είναι η μείωση της ένδυας. Θα πρέπει να δούμε πώς καταπολεμούμε την απομόνωση, πώς ε, μπορούμε να μειώσουμε τα εμπόδια οποιασδήποτε φύσεως, να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και υπάρχουν και άλλα πολυπιαστικά ζητήματα, τα περιβαλλοντικά, οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, ε, τα, οι βιώσιμοι στόχοι της χελιετίας, προβλέπουν μια α, συνεκτικότατη ατζέντα για μια αναπημένη πολιτική η οποία θεωρούν ότι αποτυπώνει το Aid for Trade. Επικεντρώνεται μεν στους οικονομικούς στόχους, από την άλλη και στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Και όπως είπε ο Μάικλ, είναι σημαντικός ο ρόλος που έχουν να παίξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο πλαίσιο του Aid for Trade. Έχει αλλάξει και το σκηνικό και το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα η ευρωπαϊκή κοινότητα θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη για να κατακτήσει μια δυναμική και φιλόδοξη πολιτική στο Aid for Trade. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν μίλησα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα σημαντικά τα σχόλια και θα πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση του χρόνου και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία στο βαθμό που μπορούμε. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση με Skype. Yes, thank you very much. Ε, okay, so, ε, Ωραία λοιπόν. Είναι μετά τα μεσάνυχτα σε σας εκεί στην Καλιφόρνια, οπότε εγώ θα σας πω καλημέρα. Χαίρομαι που δέχεστε αυτή την ε, συνδιάσκεψη μέσω Skype αυτή τη δύσκολη ώρα. Είστε η κυρία Κάτι Σουόμινεν. Θα σας παρουσιάσω στα γρήγορα και μετά θα σας δώσω το λόγο εάν αυτό δεν ε, υπάρχει, αν δεν σας δημιουργεί πρόβλημα. Um, Όπως ακούσαμε, το θέμα της αξιολόγησης ήταν η διασυνδεσιμότητα και πιστεύω πως ε, αυτό απηχεί την κατανόηση που υπάρχει στη διεθνή κοινότητα δωρητών πως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου, να ανοίξουμε δυνατότητες για όλες τις εταιρείες, τις μεγάλες και τις μικρές, να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Φίλιο. Και αυτό ανοίγει ιδιαίτερε πιθανότητες για όσους οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από το εμπόριο για πάρα πολλά χρόνια, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι γυναικείες επιχειρήσεις και οι αγροτικές ε, επιχειρήσεις γιατί online είναι πιο ορατές γιατί τους βλέπουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις από άλλα μέρη του κόσμου μέσα σε μια στιγμή. Να σας δείξω λοιπόν κάποιες διαφάνειες, να σας πω πως τις έχετε κι εσείς. Ε, θέλω να δούμε την επόμενη που είναι η δεύτερη, που είναι οι εξαγωγείς και οι πολιτές online και βλέπετε τις επιδόσεις ε, στη διαφάνεια. Εγώ συνεργάστηκα με την ε, Υπηρεσία για την Διεθνή Αναπτυξική Βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και κοιτάξαμε σε μια έρευνα πώς οι μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και πώς ε, ωφελούνται. Και ένα από τα ευρήματα που ήταν εκπληκτικά είναι όταν, όταν συγκρίνουμε με αυτούς που δεν κάνουν παρουσίες online με αυτούς που δεν κάνουν, θα δείτε πως αυτοί που δεν κάνουν online αγοροπολισίες δεν εξάγουν κιόλα. Είναι τρεις φορές λιγότερο οι δυνατότητες που έχουν για εξαγωγές. Άρα λοιπόν το 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξάγουν ε, από τις χώρες αυτές και το 60% αυτών ε, το κάνουν μέσω online δυνατοτήτων. Επίσης, για όσους κάνουν αγοραπολισίες όχι online, να σας πω πως έχουν πολύ λιγότερο διαφοροποιημένες αγοραπολισίες, ε, είναι περιορισμένες οι αγορές οι οποίες εξάγουν και αν δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν ε, ε ή πολλούν online θα δείτε πως ε, είναι πολύ πιο διαφοροποιημένες οι εξαγωγές τους σε περισσότερες αγορές ε, από ό,τι θα φανταζόμασταν. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται στο eBay ή στο Alibaba θα δείτε πως εκεί είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, δηλαδή στέλνουν σε 40 ή 50 χώρε μέσω eBay αυτέ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αν δούμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι καταπληκτικά, μπορεί ε, να πει κανεί και γιατί να ασχοληθούμε λοιπόν. Α ε, ας αφήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο να κυλήσει και θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όχι, όμω κατανοούμε πω έτσι όπω ε, και στο Aid for Trade κάναμε κάποιε σκέψει, έτσι και εδώ υπάρχει κάποιο περιβάλλον το οποίο θα πρέπει εμεί να να στηρίξουμε έτσι ώστε οι συνθήκες να είναι κατάλληλες και να αναπτυχθεί ε, αυτό το εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ψηφιακό εμπόριο είναι κάπως διαφορετικό από το παλιωμοδίτικο εμπόριο. Έχεις άλλες υποδομές, αλλά έχεις και τις δυνατότητες ε, διευκόλυνσης εμπορικής που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ιδιαίες συνθήκες, δηλαδή πληρωμές online για παράδειγμα. Ε, ε, πηγής χρηματοδότησης ε, για όσους έχουν ε, ανάγκη ε, βραχυπρόθεσμης στήριξης μέσω κεφαλαίων μέσω πιστώσεων. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές πηγαίνουν, βγαίνουν online, είδατε πως τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Γι' αυτό θα πρέπει να στηριχθούν. Εγώ είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τις επιχειρήσεις αυτές. Οκ, πείτε μου, ποια είναι τα προβλήματά σας, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιο είναι το περιβάλλον σας, σας υποστηρίζει ε, αρκετά. Δώστε 10 για το καλύτερο, 1 για το χειρότερο. Και οι περισσότεροι είπαν το περιβάλλον τους είναι 5 με 6. Δηλαδή δεν είναι ε, χαρούμενοι ε, με το περιβάλλον στο οποίο γίνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, γιατί αν δούμε τα αποτελέσματα από τον Μπαγκλαντές ή την Κάνα θα δείτε πως στις φτωχέ χώρες εκεί τα αποτελέσματα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή οι επιχειρήσεις στα στοιχεία αυτά δίνουν 2-3 βαθμούς από τους 10 που θα μπορούσαν. Και κυρίως το πρόβλημα είναι ε, τα logistics και η ε, δυνατότητα δανειοδότησης. Θα δείτε εδώ και περισσότερες λεπτομέρειες Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για όλους. Στην κορυφή θα δείτε πως είναι τα logistics και τις διασυνοριακές διεκπαιρεώσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά δυσκολεύονται και παράλληλα οι ψηφιακές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται ως εμπόδιο, ε, εμπορικό εμπόδιο. Δηλαδή, τι γίνεται ε, με την ε, εμπορική ευθύνη για παράδειγμα. Είναι διαφορετικοί οι κανόνες από αγορά σε αγορά. Είναι διαφορετικοί οι κανόνες για το copyright. Οπότε όλα αυτά τα logistics ε, τελικά δημιουργούν πρόβλημα. Αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε πως μπορεί κανείς να απαντήσει εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Οι εταιρείε πάντα κάποια παράπονα θα έχουν. Γιατί να ασχοληθούμε εμείς. Γιατί. Γιατί τα οικονομικά κέρδη είναι μεγάλα. Και από την έρευνα αυτή διαπιστώσαμε πως αν οι επιχειρήσεις ε, βλέπανε από το ηλεκτρονικό εμπόριο να φερούνται τα τρία βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, τότε θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εγχώριες ε, πωλήσει 34% και τις διεθνείς πωλήσει κατά 30%. Καταλαβαίνετε πως αυτό είναι τεράστιο για μια μικρή επιχείρηση. Εγώ έχω μια μικρή επιχείρηση δική μου και αν κάθε χρόνο κάνω μια αύξηση τη τάξη του 30% γιατί το ρυθμιστικό εμπόδιο έχει... Ε, ε ξεπεραστεί, θα ήμουν πραγματικά υπερχαρούμενη. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν και πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με το Aid for Trade. Εμείς αυτή τη στιγμή χαράσουμε πολιτική και θεωρούμε πως προσφέρει μια τεράστια ε, ευκαιρία η ψηφιοποίηση το ηλεκτρονικό εμπόριο για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκεί, αλλά χρειαζόμαστε στοιχεία και πρέπει να κάνουμε κάποιες ε, ε, να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, να οριοθετήσουμε προτεραιότητε και να δούμε πώς θα προωθήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, όπως επίσης και τι θα κάνουμε με τις θεσμού και υπηρεσίε που έχουν σκοπό την προώθηση ε, του εμπορίου. Και οι καταναλωτές ε, έχουν μπορέσει να καταλάβουν τι πεδίο ανοίγεται για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις. Στο ιδιωτικό εμπόριο έχουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληρωμής για παράδειγμα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα ποιες είναι οι προκλήσεις και οι κυβερνήσεις. Καλό θα ήταν να το συζητήσουν μαζί τους. Ε, πήγα σε χώρες όπως η Τουρκία ή το Μπαγκλαντές ή το Μεξικό και εκεί γίνεται πολύ θετικό δημόσιο διάλογο για αυτές τι πολιτικές και για τα προγράμματα τα οποία προωθούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι λοιπόν τεράστιε ευκαιρίε που προσφέρονται και θέλω να σα δείξω και την τελευταία διαφάνεια. Όταν δούμε ποιο είναι αυτό το θετικό περιβάλλον για το εμπόριο και για, το για τον ιδιωτικό κλάδο, δεν χρειάζεται εμεί να φέρουμε τα πάνω κάτω. Όχι, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τι θα γίνει με τη ρύθμιση, με τη διευκόλυνση, με το εμπορίο, με τις εξαγωγές. Είναι τα ίδια ζητήματα, απλώς έχουμε εμφιαλώσει το παλιό κρασί σε νέα μπουκάλια. Θέλουμε εδώ να κάνουμε κάποιες ε, αλλαγές έτσι ώστε να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή, να έχουμε δυνατότητες συγχρηματοδότησης κτλ. Ε, και να κάνουμε συνέργειες μεταξύ ε, για παράδειγμα των τεχνολογικών εταιριών και των ε, ε, εξαγωγικών θεσμών έτσι ώστε τα αποτελέσματα είναι θετικά για όλους. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τόσο εύστοχη παρέμβαση και τις ενδιαφέρουσες ιδέες. Να στραφώ τώρα στους συμμετέχοντες, να ευρωβουλευτές και να ζητήσω τις ερωτήσεις, τα σχόλιά σας οι τρεις ε, συμμετέχοντες στο πάτελ θα είναι εδώ για να απαντήσουν. Έχετε το λόγο, κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Επίκαιρη. Η συνάντηση των δύο επιτροπών για την ανάπτυξη και των δύο ε, οργανισμών. Καλώς ορίζω την πρωτοβουλία. Να ρωτήσω τους συμμετέχοντες, τους προσκεκλημένους μας, για τη σημασία του να υπάρχει ένα ευνοϊκό εμπορικό περιβάλλον ώστε να προσελκύονται επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης. Πώς βλέπετε τις δυνατότητες των προγραμμάτων Aid for Trade, κατά πόσον μπορεί να προωθήσουν διαφανή μάλλον να προωθήσουν τη διαφάνεια, ένα καλό νομοθετικό και κυβερνητικό περιβάλλον και την ε, καλή φορολογική πολιτική. Τι ε, δυνατότητες έχουμε εδώ να επηρεάσουμε τα πράγματα. Και όταν μιλάμε για το Aid for Trade, προφανώς μιλάμε για επιχειρήσεις και εταιρείες. Πώ βλέπετε τη λογοδοσία των εταιριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά, την προστασία των ελλαδικών δικαιωμάτων. Παίζουν και αυτά ρόλο στην αναθεώρηση του προγράμματο Aid for Trade. Είναι σημαντικά. Ευχαριστώ. Επόμενη η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ. Επίκαιρη συζήτηση όντω. Ήθελα λίγο να επικεντρωθώ στις λεπτομέρειες της ψηφιακής διάστασης και την ανάγκη πρόσβασης στο ανοιχτό ίντερνετ όταν μιλάμε για εμπόριο και ηλεκτρονικό εμπόριο. Εάν μπορούσαν λίγο οι συμμετέχοντες να μας πούν ποιο είναι το περιβάλλον που διευκολύνει τα πράγματα, συγκεκριμένα έχω κατά νου τις διασφαλιστικές δικλείδες για τα δικαιώματα των ανθρώπων στο ίντερνετ και την ασφάλεια. πώς θα είναι το περιβάλλον ευνοϊκό, πώς θα υπάρχουν απαραίτητοι νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να μην δημιουργηθούν παραθυράκια στις ψηφιακές υποδομές, παραθυράκια που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν κάποιοι εις βάρος και της κυβερνοασφάλειας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Πώς μπορούν αυτά να αποφευθούν με την ε, μόχλευση της ε, βοήθειας, της αναπτυξιακής βοήθειας και του προγράμματος Aid for Trade, ιδίω γιατί ο ιδιωτικό τομέα παίζει εδώ πολύ σημαντικό ρόλο. Δεύτερη ερώτηση. Διαφθορά. Πώς μπορεί να αποφευθεί και πόσο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επηρεάσει θετικά πράγματα στη συνεργασία με τις κυβερνήσεις των αυτοσόμενων χωρών. Τέλος, και αυτό είναι κάπως ευρύτερη παρατήρηση, αλλά πάλι ιδιαίτερη ενδιαφέροντο για μένα, βλέπουμε να διαμορφώνεται μια τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κάπω επικίνδυνη τάση πολλά εργαλεία εξωτερική πολιτική, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη και το εμπόριο, χρησιμοποιούνται ω ε, όργανα ε, για την αναχέτηση των μεταναστευτικών ροών προ την Ευρώπη. Μπορείτε να μα πείτε τι επιπτώσει έχει αυτή η τάση. Εάν η αναπτυξική βοήθεια και κατ' επέκταση και το εμπόριο γίνουν τελικά εργαλεία, όπλα για να ε, αμυνθούμε κατά της μετανάστευσης, και τι θα γίνει με την έμφυτη αυτή ανάγκη να ε, επεξεργαστούμε σωστά τους πολιτικούς μας στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Να... Μην κάνω κι εγώ λοιπόν ξεχωριστή ερώτηση, αλλά να πω ότι συμφωνώ μαζί σας. ήθελα να ρωτήσω ακριβώς για την ε, σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Ε, η κυρία Ροντρίγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη του πάνελ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπαν και για τα όσα ακούσαμε και μέσω Skype. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, για το ψηφιακό χάσμα. Δώσατε ένα νούμερο. Είπατε περίπου ε, τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα όταν οι ιδιωτικές επενδύσεις, εφόσον αυτές είναι πολύ φτωχές περιοχές, δεν θα γίνουν. Γιατί δεν υπάρχει ούτε αγοραστική αξία ε, δύναμη έτσι ώστε οι χρήστες να μπορέσουν να πιέσουν για να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Πώς θα καλύψουμε λοιπόν αυτό το ψηφιακό χάσμα και θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για να το καταπολεμήσουμε. Πώς μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση για τις απαραίτητες υποδομές. Και δεύτερον, όλοι, και συμφωνώ σε αυτό, Είπατε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ δημοσίου ε, και ιδιωτικού κλάδου, τα διάφορα ΣΔΙΤ. Έχετε κάποια... Έχετε εξετάσει πώς έχουν λειτουργήσει αυτά μέχρι σήμερα και ποιοι είναι οι μηχανισμοί που θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και δίκαιοι σε αυτές τις επενδύσεις. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη η κυρία Κιτών Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσει έχω κι εγώ. Παίρνοντα αφορμή από τι ερωτήσει τη Χέιντι για τα εργασιακά και την προβλητική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή να θεωρεί τη στρατηγική τη για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη με τα κεφάλαια για το εμπόριο στι αναπτυξιακέ συμφωνίε. Νομίζω ότι το Aid for Trade σκοπό έχει να διασυνδεθεί με του στόχου τη χιλιετία και τη σχετική ατζέντα. Ε, θα πρέπει να πάρουμε τα καλύτερα παραδείγματα του Aid for Trade για να δούμε που υπήρξαν καλές πρακτικές και που είναι ε, δυνατές οι βελτιώσεις τα εργασιακά ώστε να διασυνδεθούν με τις εμπορικές πολιτικές και τα σχετικά προγράμματα. Το ίδιο και για τα περιβαλλοντικά. Δεύτερο στοιχείο για το ψηφιακό εμπόριο. Έχω κάποιες απορίες, διότι είμαι σκιώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών για τις σχετικέ διαπραγματεύσεις εμπορικών θεμάτων ε, και διαπραγματευόμαστε όλα τα θέματα GATT σε σχέση με το ε, ψηφιακό περιβάλλον και την ε, μεγάλη ενδυνάμωση του ίντερνετ. Αυτά πηγαίνουν ε, παράλληλα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια παράλληλη πορεία και με τις συζητήσεις στο Aid for Trade, γιατί αυτή τη στιγμή βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει λόγω του παγκόσμιου σκηνικού παύση, τη διαπραγματεύση, αλλά πώς λαμβάνεται υπόψη η ψηφιακή διάσταση εδώ. γιατί θα πρέπει κάπως να τα πούμε τα πράγματα, είναι οι εμπορικές συμφωνίες με τις εμπορικές διευκολύνσεις που παρέχουν μέσω των ψηφιακών μια ευκαιρία για τις αναπτυσσόμενε χώρες ή οι υπόλοιπε συμφωνίες ΤΙΖΑ είναι ε, αυτές που θα πρέπει να προτεμηθούν. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ των δύο και θα πρέπει να τα συνδυάσουμε ίσως στο επίπεδο του Aid for Trade. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, έχουν ακόμη δύο. έχω ακόμη δύο μιλητές, αλλά θα ήθελα τώρα να κλείσω τον κατάλογο των αγορητών για να έχουμε χρόνο και για τις απαντήσεις τον κύριο Σούστα. Καταρχά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι παρουσιάσει, οι οποίε ήταν πάρα πολύ σημαντικέ και νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνουμε να συμπεριλάβουμε και την ιδιωτική ε, οικονομία σε θέματα εμπορίου αλλά και σε θέματα ανάπτυξη. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό επιτεύγμα. Για το Aid for Trade θα ήθελα να κάνω μόνο το, μία ερώτηση. Υπάρχει περιφερειακή και τοπική διαφοροποίηση. Ποιοι είναι οι παράγοντε που έχουν σημασία περιφερειακή μεταξύ δηλαδή ε, των χωρών αλλά και στο ιστορικό των χωρών γιατί φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να είναι διαφορετικές ε, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες ε, σε αστικό περιβάλλον ή στην Ήπεθρο και κατά πόσον υπάρχει και περιφερειακή, μάλλον συγγνώμη, τομεακή διαφοροποίηση μεταξύ των τομέων της οικονομίας. Κατά πόσον δηλαδή σε κάποιους τομείς είναι πιο σημαντικά κάποια μέτρα και σε κάποιους άλλους είναι λιγότερο σημαντικά. Αυτό θα με ενδιαφέρει Σα ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, τελευταία ομιλητρία, κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά με διάσταση πολύ γρήγορα αναφέρθηκε μεν, αλλά γενικώ και ορίστος. Ε, διερωτώ με, η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται διεθνώ σε σχέση με τον ΠΟΕ, τι ε, επίδραση μπορεί να έχει στο Aid for Trade. Είπατε ότι είναι θεμελιώδη ο ρόλος που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι. Σκέφτεστε ήδη τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να παίξει η κατάσταση των πολιτικών πραγμάτων Επίση, Επίσης, για το θέμα της ε, ψηφιακής διασύνδεσης. Όλοι οι προσκεκλημένοι μας είπαν ότι πρέπει να συνδυάσουμε τα διαφορετικά στοιχεία του πάζλ, ε, τις υποδομές, την ενίσχυση των ε, θεσμών και των αρμοδιοτήτων. Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερο και θα ήθελα να μπορείτε να μας αναπτύξετε περαιτέρω το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι διαφορετικοί πυλώνες της βοήθειας, αλλά ενδεχομένως και με διαφορετική συμμετοχή των κυβερνήσεων ή τέλος πάντων όσων συντονίζουν τις διάφορες απαραίτητες δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να στραφώ και πάλι στους εξαίρετους προσκεκλημένους μας. θα έχετε μια μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσετε. Θα έχετε τρία λεπτά ο καθένα. Κύριε Ρόμπερτ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αδύνατο αυτό που ζητάτε. Να θίξω κάποια από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στα σχόλια. Το επενδυτικό κλίμα. Τη δουλειά αυτή βεβαίω την κάνουμε οπωσδήποτε για την πρωτοβουλία Aid Trade και την εκπόνησή τη. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις που συζητούνται αυτή τη στιγμή στον ΠΟΕ σε σχέση με τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Θα γνωρίζετε τη Συμφωνία Διευκόλυνσης του Εμπορίου Αλλά έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιου μήνε οι συζητήσεις μεταξύ των μελών για το πώς να βελτιώσουμε το επενδυτικό κλίμα. Αυτά θα συζητηθούν και τους ερχόμενους μήνες, όπως θα πλησιάζουμε στην 11η Σύνοδο του Buenos Εδώ ένα θέμα λοιπόν που ακούστηκε επίση είναι η λογοδοσία. Οι συζητήσει περί διαφθορα Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι συμφωνίε διευκολυνση των εμπορίου όχι απλώ προσφέρουν προβληψιμότητα σε σχέση με αυτέ τι διαδικασίε. Και εδώ έχω κατά νου τη συμφωνία του, την σημασία του τελωνιακού εισοδήματο, των τελωνιακών εσόδων για ένα μεγάλο αριθμό αναπτυσσόμενων χωρών για τα δημοσιονομικά τους. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί προβλεψιμότητα και δυνατότητα ε, απόκτησης εσόδων ε, και αν προσθέσουμε εδώ την ψηφιακή διάσταση και με κάποια παραδείγματα που χρησιμοποιήσαμε στην διαδικασία για την παγκόσμια αναθεώρηση του ΕΦΟΤΕ, είδαμε πω η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά, να αυξήσει το εισόδημα τη κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια, ένα σκέλο σημαντικό που πάλι έχει να κάνει με το ψηφιακό περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, και αυτό το κομμάτι, νομίζω, ε, εμείς πιο πολύ έχουμε στραφεί στις συζητήσεις μας τα πρώτα βήματα. Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες ε, ήδη ε, είναι στα πρώτα βήματα. Δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο της ασφάλειας να συζητιέται στο σημερινό στάδιο σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Είναι σημαντικό και ενδιαφέρον και στρέφομαι πάλι στις συμφωνίες διευκόλυνσης των πορείων είναι ότι μπορεί να υπάρχουν οικονομικές συνέπειε για τη μετανάστευση, αλλά και φυσικές ε, καταστροφές, ενδεχομένως ε, καιρικέ μεταβολές που να ε, αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Άλλο αίτιο μετανάστευσης και αυτό. Εδώ κάτι σημαντικό που ακούστηκε στη συζήτηση και στις δικές μας συζητήσεις είναι πως οι αποτυχημένες τελειωνικές διαδικασίες μπορεί να δημιουργήσουν αυξημένες ανθρωπιστικές πιέσεις. Το να ευθυγραμμιστούν λοιπόν οι τελειωνιακές διαδικασίες και να μειωθούν οι καθυστερήσεις, να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης, μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να μείνουν και να χτίσουν τις ζωές τους αλλού. Ε, το εργασιακό περιβάλλον, ε, τα σχετικά θέματα. βεβαίω αυτά στους στόχου της χιλιετία καλύπτονται. Όλα τα μέλη του που έχουν προσυπογράψει στις σχετικές απαιτήσει των στόχων της χιλιετία. Και υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς ε, κάποια μέλη του ΠΟΕ θα ήθελαν να ε, επιλύσουν το θέμα αυτό. Κάποιοι θέλουν διμερείς σχέσεις και συμφωνίες, κάποιοι άλλοι πολυμερείς ή τέλος πάντων έχουν άλλη προτίμηση και εδώ καθεξής. Τέλος, Πρόεδρε, για το αν θα υπάρξουν ξεχωριστοί κανόνες μέσω των συμφωνιών ΤΕΦΤΙΣΑ και για ποιες χώρες ή διατάξεις ε, προτιμησιακές για τις φτωχότερες χώρες. ή συζητήσεις έχουν πολύ δυναμικό χαρακτήρα στον ΠΟΕ. Τα πράγματα αλλάζουν διαρκώς και ε, με την διευκόλυνση των επενδύσεων και το e-commerce, το ηλεκτρονικό, πρόγραμμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το σχετικό πρόγραμμα, ταυτόχρονα μας απασχολούν και θέματα όπως η διευκόλυνση των, ε, της παροχής υπηρεσιών, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή η μετανάστευση. Δηλαδή, η συζήτηση είναι κάποιος, κάπως πιο ευρεία από ό,τι μπορεί να έχετε σκεφτεί. Νομίζω ότι εξήγησα τα τρία λεπτά και τα ξεπέρασα κιόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να στραφώ τώρα στον ε, δεύτερο προσκεκλημένο μα. Προσκεκλημένο μα. Sorry. I will also focus on a few points and I'm not able to end. Σα ευχαριστώ πολύ. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να απαντήσω όλε τι ερωτήσει. Το θέμα τη μετανάστευση νομίζω ότι ήταν ο πρόεδρο του Μέξικο που στη διαπραγματεύσει για την ΑΦΤΑ είπε ότι κοιτάξτε, είτε προϊόντα θα σα στείλω, είτε ανθρώπου θα σα στείλω. Τώρα τα πράγματα φυσικά έχουν δυσκολέψει λίγο, αλλά είναι δύσκολο να υπάρχουν πραγματικά βιώσιμε προοπτικέ οικονομική ανάπτυξη για τον κόσμο. Και αυτό είναι το στοιχείο που πραγματικά αποτρέπει τη μετανάστευση. Ένα από τα στοιχεία. Ένας από, μάλλον, τι προϋποθέσεις, μία από τις προϋποθέσεις για να υπάρξει σωστό οικονομικό κλίμα είναι να υπάρχει σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο και χρειάζεται λοιπόν τεχνική αρρωγή ε, συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει τέτοιες συστάσεις βάσει και του παραδείγματος της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο διαδίκτυο. 500 εκατομμύρια το χρόνο δαπανώνται. Αυτό δεν ακούγεται πολύ μεγάλο ποσό, αλλά αυτό είναι για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και να σας πούμε ότι αυτό έχει να κάνει και με τις τιμές. Εξετάσαμε για παράδειγμα κατά πόσον υπάρχει συμμετοχή ιδιαίτερη του ιδιωτικού κλάδου σε χρηματοδότηση δύο ετών και κατά πόσον υπάρχει μόχλευση 200 δισεκατομμύρια ήταν αυτή η δυτική μου όχλευση. Έχει να κάνει αυτή με την κοινωνική ευθύνη. Έχει να κάνει. Πιστεύω ότι όλο και πιο πολύ ο ιδιωτικό τομέα ε, δαπανά στην ε, εταιρική ευθύνη, στην ε, κοινωνική ευθύνη. Όχι γιατί προβλέπεται από τους εθνικέ προδιαγραφέ, αλλά επειδή είναι προ το συμφέρον τους. Το για παράδειγμα, ε, μία σειρά κρατών συγκεντρώθηκαν και μίλησαν με εταιρείε και με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ για να βελτιώσουν τι συνθήκε στα εργοστάσια και οι αξιολογήσει καταδεικνύουν ότι διαπιστώνονται και οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση και έτσι βλέπουμε ότι μπορούμε να ενταχθούμε από την κάθε περίπτωση. Έχουμε το Παγκοσμίο Οικονομικό Φόρουμ, έχουμε και τις διεθνεί οργανώσεις στην Γενέβη. Γίνεται καλή δουλειά και ξέρουμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει σε συνεργασία με τον δημόσιο και τον κλάδο. Τώρα, πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι η βοήθεια είναι καλή πραγματικά και έχει καλά αποτελέσματα. Θετικά. Ο ΑΣΑ θεωρώ ότι έχει καταρτήσει μια εξαιρετική, αν θέλετε, ένα εξαιρετικό κατάλογο προδιαγραφών σε ό,τι αφορά το κατά πόσο είναι θετικό αντίκτυπο, σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων, την προώθηση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν αποδεχτεί μετά από χρόνια συνεργασία. Εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Και τέλο, να σα πω ότι όταν παρευρεθήκα στην Γενέβη και συζητήσαμε την συμμετοχή του ιδιωτικού κλάδου, κάποια κρατημέλη επανέλαβαν αυτές τις αρχές του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της αρρωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να συμπεριληφθεί ο ιδιωτικός κλάδος και όπως ξέρετε η συμμετοχή του ιδιωτικού κλάδου δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένα τον Ολλανδικό, Φιλανδικό ε, ιδιωτικό κλάδο έχει να κάνει με την ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας στις χώρες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί οι αρχέ μα και οι προτεραιότητέ μα δεν είναι αυτέ που ήταν πριν από 20-30 χρόνια που θέλαμε να προωθήσουμε απλά τι δικέ μα επιχειρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο, και ελπίζω να έχουμε ακόμα σύνδεση με Los Angeles. Ναι, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέσσερα σχόλια επιτρέψτε μου για τι κριτικέ αυτέ ερωτήσει. Πρώτο σχόλιο που έγινε για το ρυθμιστικό περιβάλλον. Κάτι που έμαθα στη διάρκεια της ε, ανάλυσης αυτής για τις προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι όντως όλα αυτά τα ζητήματα, όλοι αυτοί, όλες αυτές οι ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις έχουν ε, μεγάλη σημασία και για τις μικρές επιχειρήσεις που ε, δραστηριοποιούνται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουμε πολλές προκλήσεις λοιπόν να αντιμετωπίσουμε. Ένα μεγάλο περιθώριο ευκαιρίας ανοίγει τώρα, μιας και τόσες πολλές χώρες κινούνται προς την ανάπτυξη των μικρομεσαίων τους επιχειρήσεων προκειμένου να μετακινηθούν στο διαδίκτυο. Εδώ θα πρέπει να γίνει λοιπόν η τομή. Είναι καλή η ορμή που υπάρχει τώρα, το κλίμα που υπάρχει τώρα, για να δείξουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες ότι κοιτάξτε, θέλετε πιο πολλές εξαγωγές, πιο πολύ ε, εμπόριο στο διαδικτύο, αναπτύξτε αυτό το σκέλος της επιχειρηματικότητας και αξιοποιήστε την ευκαιρία για να ε, κάνετε κάποιες μεταρρυθμίσεις φορολογικές και ρυθμιστικές. Αυτό έχει να κάνει και με τα θέματα μετανάστευσης. Έχω συνεργαστεί με επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, μικρές και μεγάλες αναπτυσσόμενες ε, χώρες και σε μεγάλες ε, χώρες, τεράστιες αγορές τίθεται το θέμα των όρων εισαγωγή ό,τι αφορά τα προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα, δεν θέλω να αμφισβητήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν ερωτήματα σε ό,τι αφορά τι αντισώμενε χώρε. Ε, ζητούν ε, υψηλότερα πρότυπα την σε ό,τι αφορά την πώληση προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά γιατί υπάρχουν ε, πραγματικά τελωνιακές, ε, τελωνιακά εμπόδια, φορολογικά εμπόδια, σε ό,τι αφορά προϊόντα μικρή αξία. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την πρόσβαση τέτοιων ε, χωρών, χωρών στις ευρωπαϊκές αγορές και σε άλλες αγορές όπου τα όρια δεν ήταν πολύ χαμηλά. Ένα τρίτο ζήτημα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό είναι τα θέματα προστασίας του καταναλωτή. Θα πρέπει να τα κοιτάξουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως ξέρετε, είναι τόσες πολλές οι δραστηριότητε ε, που λαμβάνουν χώρα στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη μεταρρύθμιση και του ρυθμιστικού πλαισίου για την προετοιμασία για την ψηφιακό περιβάλλον και είχα μια ευκαιρία να κάνουμε μια σχετική ανάλυση στη Λατινική Αμερική και είδα πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρε για να εισαγάγουν κανονισμού για την νόμικη ευθύνη, για την προστασία των καταναλωτή, την προστασία των επιγραμμικών πωλήσεων. Και παράλληλα, όταν μιλάμε τι επιχειρήσει, εκφράζεται η ανησυχία ότι σε κάποιε περιπτώσει οι κυβερνήσει τα πράττουν αυτά λίγο απομονωμένα στι αναπτυσσόμενε χώρε. Καταπίζουν δηλαδή τι πολιτικέ του και δεν τι ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενσωματώσουν τι ανάγκε ε, των ε, μικρών επιχειρήσεων. Το να υπάρχει λοιπόν ένα διάλογο για να καταρτιστεί τελικά ένα ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο και να μην είναι υπερβολικές, υπερβολικοί περιορισμοί για το ψηφιακό εμπόριο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτή οδός επικοινωνίας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου κλάδου. Προκειμένου και ο ιδιωτικός κλάδος να εκφράσει τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του στο πλαίσιο αυτό. Κάποια παραδείγματα με ανησυχούν, γιατί φαίνεται ότι γίνεται κάπως ε, μονόδρομα, χωρίς επαφή με τον ιδιωτικό κλάδο. Τέταρτος, ε, τέταρτο θέμα, σε ό,τι αφορά και τα σχόλια από Ισπανία, σε ό,τι αφορά δηλαδή στην πράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το πώς ε, εφαρμόσονται στην πράξη. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, ενδείξεις για το τι γίνεται από τις νομικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, στο Μπουρούντι, στην Αφρική, για επενδύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε το τι έγινε και πριν από τρία χρόνια, αλλά με τρεις ε, τρόπους θα πρέπει να κοιτάξουμε τις συμπράξεις αυτές. Καταρχάς, τον διάλογο στις αναπτυσσόμενες χώρες φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλο χάσμα μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου κλάδου σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την κατανόηση της τεχνολογίας και των κανονισμών που χρειάζονται προκειμένου οι τεχνολογίες πραγματικά να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις και τον καταναλωτή φυσικά στη τελική ανάλυση. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν ιδιαίτερα το δημόσιο κλάδο ποιες είναι οι ανάγκες και οι προκλήσεις του ιδιωτικού τομέα Νομίζω ότι αυτό θα δώσει πολύ καλές ευκαιρίες. Δεύτερο ζήτημα, να μιλήσουμε για νέες εταιρικέ ε, σχέσεις. Ε, για παράδειγμα, οι πελάτες φαίνεται ότι ανησυχούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διάδοση των μικρών πακέτων σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν στην τελική ανάλυση τι περιλαμβάνουν αυτά τα μικρά πακέτα, δεν μπορούν να τα παρακολουθούν ε, και να τα ανεχνεύουν. Μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια καινούργια δεδομένα προκειμένου να υπάρχουν online πλατφόρμες για να γίνει αξιολόγηση του κινδύνου. Να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα αυτά. Προκειμένου να ξέρουμε όλα αυτά τα πακέτα που αποστέλλονται, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο. Να καταχωρούνται. Και τελευταίο στοιχείο, συγχρηματοδότηση. και για εσωτερική κατανάλωση αλλά και για εξαγωγές στην ψηφιακή εποχή. Τέτοιες δραστηριότητε δεν μπορούν να γίνουν μόνο από τον ε, ιδιωτικό, από το δημόσιο κλάδο. Θα πρέπει να συμμετέχει και ο ιδιωτικό. Δεν αρκεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος από μόνο του. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συμμετάσχουν για να υπάρξει χρησιμοποιηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε όλα αυτά στα πλαίσια του Aid for Trade. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Ευχαριστούμε όλους τους πανελίστες για την πολύ καλές, πολύ καλές παρεμβάσεις. Πολλές καλές ιδέες ακούσαμε και πολλά εύστοχα συμπεράσματα. Έτσι ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο πάνελ και νομίζω ότι πάρα αυτά θα αλλάξουμε τη σύνθεση του πάνελ. Και με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη μου χαρά θα δώσω την προεδρία στο δεύτερο τμήμα αυτού του πάνελ στον συνάδελφο κύριο Βαράινεν. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα κάνατε στο κομμάτι του της ακρόασης που σας αντιστοιχούσε. Έχουμε καθυστερήσει κάπως. Νομίζω πάντως πως παρόλα αυτά δίκιο θα ήταν να δώσουμε στους ε, συμμετέχοντες στο πάνελ τον χρόνο που είχαμε προβλέψει, που είναι τα 8 λεπτά. Αν βέβαια μπορείτε να τα πείτε πιο γρήγορα, καλό θα ήταν. και βλέπω ότι έρχεστε για να καθίσετε. Όσο λοιπόν σας περιμένουμε, εγώ θα ξεκινήσω με τα εισαγωγικά μου σχόλια. Speaker Σήμερα έχουμε τον κύριο Γιάγκερ που είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναπληρωτής Διευθυντής στην ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Είναι μία συνάδελφος που, που εργάζεται από το 2005 ε, στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη ξεκίνησε ως αρμόδια για θέματα ενέργειας στην Γενική Διεύθυνση στην Ενέργειας και ε, Συγκοινωνιών. Ήταν κάποτε και διευθύντρια του ε, γραφείου του Αρμόδιου Επιτρόπου για την Ενέργεια και έχει τουλάχιστον 10 χρόνια που εργάστηκε για την προσχώρηση της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν η πρώτη ε, πρέσβης της Σλοβενίας στην Κορεπέρ. Ε, αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Έχετε 8 λεπτά, αλλά αν μπορείτε να το πείτε και πιο γρήγορα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι Επιτροπέ για την ευκαιρία που μα δίνουν ε, να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, το Aid for Trade, έφτασε την κατάλληλη στιγμή η ακρόαση αυτή. Σα συγχαίρω λοιπόν για την οργάνωση και όπω είπα και προηγουμένω θα πρέπει να αρατηθούμε. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε το κατά πόσο το aid for trade και αν είναι κατάλληλο. Ο Επίτροπος κ. Μίμητσα είπε καμία χώρα δεν κατάφερε να πληχθεί χωρίς εμπόριο. Άρα λοιπόν το aid for trade είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που βοηθά στις χώρες να ξεπεράσουν τη φτώχεια και τις, ε, τα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να ωφεληθούν από το διεθνές εμπόριο. Το 2007 εγκρίθηκε αυτή η στρατηγική και έκτοτε τα ποσά έχουν αυξηθεί κατά 85% 13 εκατομμύρια το 2015 και είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχο ε, ταμείο παγκοσμίω. Ε, σας εξήγησα προηγουμένω ποιο κομμάτι, τι μερίδιο έχουμε στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο και παρόλα αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα πρέπει να σας πω ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Μεγαλύτερη ε, απελευθέρωση έχει αφήσει πολύ κόσμο ε, εκτός παιχνιδιού. Δεν έχουν μοιραστεί τα κέρδη ισότιμα και δεν έχουν ωφεληθεί όλες οι περιφέρειες το ίδιο. Κυρίως για όσους δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του εμπορίου και του ανταγωνισμού. Μεγάλες προκλήσεις λοιπόν έτσι ώστε να απαλληφθούν οι αρνητικές ε, επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Ξέρετε τι σημαίνει με το κλίμα, με την ισότητα των φύλων, με τις ευκαιρίες, με την παιδεία. Οπότε υπάρχει πολύ περισσότερη ανισότητα, ένα μεγάλο πρόβλημα και πάνω από τα τρία τέταρτα των ανθρώπων στις χώρες ε, εταίρους αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν επίπεδα ανισότητας υψηλότερα από αυτά τα οποία αντιμετωπίζαμε πριν από 20 χρόνια. Για το 2015 στις 48 λιγότερες αναπτυγμένες χώρες πρέπει να σα πω ότι είχαν μερίδιο κάτω του 1% στο παγκόσμιο εμπόριο και εξαγωγές και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό σχετίζονται πολύ συχνά στην έλλειψη βιομηχανοποίησης, περιφερειοποίησης, διαφοροποίησης των οικονομιών, της ε, εξάρτησης από ε, πρώτες ύλες και μη προστιθέμενη εξία από άλλες υπηρεσίες. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια κινητοποίηση με κάποιους μηχανισμούς που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Χρειάζεται λοιπόν εκεί τα ωφέλη να τα ε, στηρίξουμε έτσι ώστε με το εμπόριο να στοχευθούν οι παραγωγικές επενδύσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα μήνυμα λοιπόν για σας, η βιωσιμότητα η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα των δράσεων που θα κάνουμε υπέρ του εμπορίου και των επενδύσεων. Και όπως είπα και προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πολύ ε, φιλόδοξο ε, σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων και χάρη στις δικές σας προσπάθειες και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου θα το δημοσιεύσουμε. Έτσι λοιπόν 28 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη στρατηγική μας προς ανακοίνωση, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα κάνουμε με το Aid for Trade και είναι ακόμα κατάλληλο για τους στόχους που εξυπηρετεί. Αντιμετωπίζει The view of uh, uh, and Θα βοηθήσει στο να προωθήσουμε και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι ε, αξιοπρεπείς. Αυτά λοιπόν ε, πρέπει να τα βάλουμε στο θεματολόγιο μας, να ευθυγραμμιστούμε γενικότερα με το εμπόριο και να δούμε τι γίνεται ε, με τους στόχους χιλιετίας. Πώς μπορούμε να τους συνδέσουμε καλύτερα με τα εργαλεία που έχουμε. Και να σας πω πως από τότε που εμείς εγκρίναμε το θεματολόγιο του 2030 έχουμε προσπαθήσει να βρούμε συνένεση στην Ευρώπη. Ε, και αυτό αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να δράσουμε με τον τρόπο που θα καλύψει όλες τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Τα μισά θα τα αφήσω εκτός για να προλάβετε να μου κάνετε και ερωτήσεις, αλλά να σας πω ότι μετά τη συνένεση που επιτύχαμε, οι στόχοι μας για να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατόν θετική επίπτωση του Aid for Trade, εξασφαλίζοντας παράλληλα πως το εμπόριο θα είναι ένα πιο κατάλληλο εργαλείο και πιο πετυχημένο εργαλείο για ένα ευνοϊκό εμπορικό ε, περιβάλλον θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε περισσότερα παραδοτέα με καλύτερο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι το Aid for Trade να το χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που θα επιτρέψει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνέργειες. Πώς? Τι θα επιθυμούσαμε? Θέλουμε καταρχήν να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό και στη συνεργασία να προωθήσουμε ολοκληρωμένες και διαφοροποιημένες αποκρίσεις. Να παραδώσουμε αυτά που είναι απαραίτητα μέσω του Aid for Trade, με πιο συστηματική διασυνδεσιμότητα μεταξύ των βασικών ε, παικτών και νομίζω πως τα εργαλεία πολιτικής όπως οι εμπορικέ συμφωνίες, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι συγχωνευμένοι ε, προϋπολογισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με καλύτερο τρόπο. Και καλό θα ήταν να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα ε, των εμπορικών μας εργαλείων. Αυτή τη στιγμή είναι 39 οι αναπτυσσόμενες χώρες που καλύπτονται από τέτοιου είδους εμπορικές 93 συγγνώμη, που καλύπτονται από τέτοιου είδους συμφωνίες και οι 90 από αυτές έχουν και τη δυνατότητα του Aid for Trade. Οπότε νομίζω πως καλό θα ήταν να δούμε και τι μπορούμε να ανοίξουμε στον ιδιωτικό κλάδο, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων και να δούμε τι νέες ευκαιρίες έχουμε εκεί. Θα πρέπει, θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι νέες συνθήκες ποια είναι η νέα εμπορική πραγματικότητα, πώς μπορούμε βιώσιμη ανάπτυξη, ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη να την επιτύχουμε, να έχουμε το ηθικό και το δίκαιο εμπόριο και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις κυβερνήσεις, να είναι πιο υπεύθυνη η ε, αλυσίδα ε, ανεφοδιασμού και τέλος θα πρέπει να εξειδικεύσουμε αναχώρα εταίρο με έναν τρόπο που θα μας κάνει πιο επιχειρησιακό, πιο αποτελεσματικό, με καλύτερη παρακολούθηση και με καλύτερες αναφορές. Να σας πω πως αυτές οι προσπάθειες blending που κάνουμε δεν βρίσκονται στην έκθεση ε, του Aid for Trade, παρόλο που το 90% της μόχλευσης των, επενδύσεων, των μοχλευμένων επενδύσεων όντως σχετίζονται με το Aid for Trade. Οπότε καλύτερη ποιότητα και μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα κλίμακας και να βελτιώσουμε και την απασχόληση και το εμπόριο. Τέλος, τι είναι το Aid for Trade. Είναι μια βοήθεια για ε, καλές συνθήκες εργασίας, για αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης και για βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε. Δεύτερος ομιλητής, ο κύριος Ζίκφιτ Λέφλερ. Είναι διευθυντής της αντιπροσωπείας GITS στις Βρυξέλλες, την γερμανική ε, εταιρεία ε, για τις ε, διεθνείς κοινοπραξίες και πριν μεταφερθεί στις Βρυξέλλες το 2016 και εργαστεί στην αντιπροσωπεία GITS ο κύριος Λέφλερ εργάστηκε από το 2011 έως 2016 ε, μετά από 15 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε διεθνείς κοινοπραξίες με επαγγελματική εμπειρία κυρίως στη Μέση Ανατολή. Κύριε Λέφλερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ το INTA και την Επιτροπή σας που οργάνωσαν αυτήν την Επιτροπή και που κάλεσαν την GIDS ως μία από τις βασικές εταιρείες για τα θέματα αυτά. Το εμπόριο, κυρίες και κύριοι, πραγματικά μπορεί να είναι κινητήριος δύναμη για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Το πλήρες δυναμικό του όμως απαιτεί να αντιμετωπιστούν προκλήσεις για τους ενδιαφερομένους σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Τώρα θέλουμε να σταθμίσουμε το τι έχει συμβεί ως τώρα και τα διδάγματά μας θα είναι ζωτική σημασίας για να βελτιώσουμε την υλοποίηση των ε, ε, νέων στόχων. Η Gates διευκολύνει τη συνεργασία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου της Γερμανίας για την Ανάπτυξη και την ε, και Βοήθεια και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, κοιτάζει επιτόπου τι γίνεται ώστε να υλοποιούμε καλύτερα τις σχετικές μας πολιτικές. Τα πορίσματά μας διατίθενται στους πολιτικούς, πολιτικούς ηθήνοντες στην Ευρώπη και στις ε, συνεργαζόμενες χώρες και ενημερώνουμε για τις προκλήσεις, τους παράγοντες επιτυχίας και επιδιώκουμε το κατάλληλο μείγμα πολιτικής για να παίξει καλύτερη ε, εμπορική πολιτική για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πριν σταθώ στι προκλήσει, να σα μιλήσω για τη γερμανική στρατηγική του A4T, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017 που ονομάζεται Ελεύθερο ε, και Δίκαιο Εμπόριο για την Ανάπτυξη. Με στόχο την ατζέντα του 2030 και του στόχου τη χιλιετία, κοιτάζουμε τι διευκολύνσει για το εμπόριο ε, και την, ε, το σωστό εμπορικό περιβάλλον. Οπότε που ξεκίνησε η πρωτοβουλία, βλέπουμε κάποια ανταλλάγματα και μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών. Τονίσαμε την σημασία του πολυμερούς διαλόγου για σκοπούς πολιτικής συνοχής και προκειμένου να μην μείνει κανείς στην ε, εκτός αυτής της διαδικασίας την εκρίζωση της φτώχειας. Μαζί με άλλες γερμανικές, ε, γερμανικούς φορείς και με την συνεργασία του Υπουργείου ορίσαμε γερμανικές προτεραιότητες για τις παρεμβάσεις μας. Έτσι η νέα γερμανική στρατηγική για την ε, εμπορική στήριξη εντοπίζει έξι κυρίους τομείς. Πρώτα απ' όλα την περιφερειακή και γεωγραφική ε, ολοκλήρωση με τη σωστή υλοποίηση των διεθνών συμφωνιών. Έπειτα την εμπορική διευκόλυνση μετά τις πολιτικές υποδομές Τέταρτον, την οικονομικέ τις οικονομικές υποδομές. Πέμπτον, τις δυνατότητες παραγωγής και βιώσιμες αλυσίδες παραγωγής. Και έκτο, την, ε, τις επενδύσεις που να στρέφονται προς την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό. Μετά από διεξοδική ανάλυση των αναγκών των εταίρων μας και των διδαγμάτων που αντλήσαμε, η Γκίτς όρισε ε, μια στρατηγική για το διασυνοριακό εμπόριο. Αυτό με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων όπως ε, πολιτική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, υποστήριξη στην οικοδόμηση θεσμών ε, ανθρωπίνων πόρων και δυναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στην καρδιά των συζητήσεών μας, στο, κέντρο των συζητησιών μας, προκειμένου να πετύχουμε ε, σωστά αποτελέσματα. Οι πολιτικές μας προϊόντες είναι της ίδιας σημασίας, γιατί καλούμε τις κυβερνήσεις και τους εταίρους μας να σεβαστούν τις αρχές που έχουμε ορίσει και να τις διαδώσουν περαιτέρω. Επιπλέον, ε, θέλουμε να υπάρχουν ε, ισχυρέ σχέσει συνεργασία με εσά, ευρωβουλευτέ και άλλου πολιτικού ευθύνοντε για να υποστηριχθεί το σχετικό πλαίσιο. Τα μέτρα μα μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο αν υπάρχουν κατάλληλε πολιτικέ για να τη στηρίξουν. Θέλουμε λοιπόν να παραμείνουμε ανοιχτοί σε διάλογο με ε, εμπορικέ πολιτικέ που να έχουν γνώμονα την ανάπτυξη. Το κατάλληλο πλαίσιο και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ε, όπως τονίστηκε από τους προαλληλισσαντές, ε, με την ημερήσια διατάξη της ε, Αντισαμπέμπα και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλα αυτά επιδιώκουν ενισχυμένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Η δική μα δουλειά στην Κίτσα ε, έχει να κάνει ε, από την εμπορική πρόθεση και την ανάπτυξη του εμπορικού τομέα με τη διευκολύνση και τα εμπόρια, τι οικονομικέ υποδομέ, την πρόθεση των επενδύσεων και τη συμβουλευτική για εμπορικές πολιτικές. Αυτή η πείρα με την ε, υλοποίηση του IFT, του, ε, του Δίκαιου Εμπορίου, μας επιτρέπουν να έχουμε ε, κάποιους παράγοντες επιτυχίας που όμως αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες επιτόπου. Πρώτα απ' όλα η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και στην υλοποίηση αλλά και στη χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικό τομέα σε αυτή την περίπτωση όχι απλώ ε, αυξάνει τι δυνατότητε επιτυχία των σχετικών μέτρων, αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο για το σχεδιασμό και την ε, σωστή εκπόνηση των μέτρων αυτών. Ε, για παράδειγμα, εκ μέρου τη γερμανική κυβέρνηση, η GITS είναι μέρο τη Διεθνού Ένωση για τι Εμπορικέ Διευκολύνσει και συντονίζεται τη Γερμανική Συμμαχία για τι Εμπορικέ Διευκολύνσει στι αναπτυσσόμενε χώρε. Κάτι που συμπληρώνει τις προηγούμενες πρωτοβουλίες μας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των δύο αυτών ενώσεων είναι η στενή συνεργασία διεθνώς γερμανικών εταιριών, ώστε να εντοπιστούν ε, ε, σημεία συγχώνευσης, ε, συμφόρηση μάλλον, για τις εμπορικές διευκολύνσεις. Έτσι, χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα όπου μπορεί να συμβάλλει αυτό. Αυτέ οι ενδεχόμενε περιοχέ παρέμβαση ελέγχονται διπλά, με διασταυρώνονται με τι κυβερνητικέ προτεραιότητε και τι τοπικέ ανάγκε, ώστε ο διάλογος αυτός να οδηγεί σε συγκεκριμένα προγράμματα για την εκπόνησή τους, προγράμματα τα οποία να είναι σφαιρικά. Επιπλέον οι εταιρείε προσφέρουν την τεχνογνωσία τους και διαρκώς λειτουργούν ως ένα ε, συμβούλιο ελέγχου για το πώς προχωρούν τα προγράμματα και πώς υλοποιούνται. Τέλος, είναι λιγότερο επαχθείς ε, και ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες εξαγωγών. Ένα παράδειγμα, το Μαυροβούνιο. Ο στόχος ήταν να αυξήσουμε τον αριθμό των συγκεκριμένων αποστολών που ε, ε, περνούν από τα τελωνία σε μία ώρα από 25% σε 65%. Έτσι τα δεδομένα ε, θα, θα γίνονταν αντικείμενα επεξεργασία γρηγορότερα. Φτάσαμε ήδη το ποσοστό του 55%. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει του Μαυροβουνίου που εξαρτώνταν από την άμεση παράδοση ανταλλακτικών ιατρικών προϊόντων και το καθεξής μπορούν να εργαστούν καλύτερα. Όλα αυτά και με ανάλογα μέτρα ευθύ σε ε, άλλους τομείς. Για την ώρα έχουμε εκατοντάδε ε, συμφωνίε ιδιωτικού δημόσιου τομέα παγκοσμίω και θέλουμε να υπάρξει συνεργασία με όλου του τομεί. Είναι σημαντικό παράγοντα επιτυχία αυτό για να έχουμε υποδομέ για το εμπόριο. Δεύτερον, θέλω να αναφέρω την προώθηση τη καλή κυβέρνηση και τη διαφάνεια προκειμένου να μειωθεί το κόστο για το εμπόριο σε ένα πρόγραμμα που υλοποίησαμε στην Κεντρική Ασία και που αφορά τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Ουσπεκιστάν, το, Καζακστάν, την Κυργιζία και το Τατζικιστάν, για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον με κατάλληλες δομές για τις περιφερειακές ανάγκες ε, φροντίσαμε να τονώσουμε το διεθνές εμπόριο με τη συνεργασία πολλών κυβερνητικών φορέων σε αυτές τις χώρες και στα γειτονικά κράτη, ώστε να έχουμε ταχύτερο ε, πολυμερή διάλογο όλων των ενδιαφερομένων και να υπάρξει ανάληψη ευθύνη από όλους τους ενδιαφερομένους. Ε, προβλέψαμε μια νέα θηρίδα one-stop shop σε όλε αυτέ τι χώρε για τι θελονικές διαδικασίε και αυτή η συστηματική ανταλλαγή δεδομένων αύξηση την ταχύτητα του εμπορίου και την διαφάνεια. Η σημασία του ευνοϊκού αυτού περιβαλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι κάτι το γνωστό η ευθυγράμμιση των τελωνιακών διαδικασιών και η συμπερίληψη πολλών παραγόντων για την εμπορική επιτυχία είναι σημαντικά. Η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι βασικέ αρχέ για τη σωστή υλοποίηση τη ατζέντα του 2030. Όπω έδειξε η πείρα μα, κάποιε φορέ η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να επιτρέψει στου πολιτικού ευθύνοντε να ε, εντοπίσουν ανάγκε για πολιτική δράση. Τρίτον, η ατζέντα του 2030 στην προτεραιότητα της ε, ε, Συνολική ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνει όλους είναι μια αρχή που καθοδηγεί τη δράση μα. Ένα παράδειγμα ήταν η προώθηση των κοινωνικών και προεβαλλοντικών προτύπων στον Μπαγκλαντέ, ε, ειδικά στι εταιρείε που λειτουργούν και στην κλωστοϊφαλουργία, μαζί με, την, ε, με το Οργανισμό Εργασία και με επιθεωρητέ, ελέγξαμε τους ε, ε, εργαζόμενους σε διτεχνίες φασματών και ενδυματών για να δούμε κατά πόσο να συμμορφώνονται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Το πρόγραμμα πέτυχε τα συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα για να ονομάσω μερικά πάνω από 780 εργαστάσια, βελτίωσαν τη συμμόρφωσή τους με τους με τους διεθνείς κανόνες 500 ε, middle managers ε, βελτίωσαν την εκπαίδευσή τους και έλαβαν ειδικέ εξειδικευμένες θέσεις εργασία, ε, με τη συμπερίληψη ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στο εμπόριο. Δεν είναι μόνο πηγή οικονομικής ανάπτυξης κατά την εμπειρία μας, αλλά είναι και μια δύναμη για την βιώσιμη και σφαιρική συμπερίληψη όλων στην οικονομική ανάπτυξη και θα ε, επιταχύνω. Τελευταίο, η πληροφορήση και η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. Το εμπόριο είναι ένα διατομιακό θέμα που συμπεριλαμβάνει πολλού εταίρου. Όλοι έχουν διαφορετικέ αντιλήψει, συμφέροντα και διαφορετικού ρόλου. Πολλοί από αυτού ε, στι συνεργαζόμενε χώρε χρειάζονται την οικοδόμηση δυνατοτήτων για να υπάρξει διάδραση στοχευμένη στα αποτελέσματα και καλύτερε διαβουλεύσει ε, και διαπραγματεύσει. Αυτή την προσέγγιση την επιδιώκουμε σε όλε μα τι προσπάθειε, ώστε να να συνεργαστούν σωστά οι εταίροι και να πετύχουν να κάνουν καλή δουλειά για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Εάν θέλετε να ξέρετε περισσότερο για την αποτελεσματικότητα ή τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε στην συνδυασμό αναπτυξιακή πολιτική και εμπορίου, μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα παραδείγματα από χώρε ή των ε, οργανισμών που εφαρμόζουν όσα έχουμε σκεφτεί. Ε, δείτε τον ιστοτόπο τη ακρόαση, αν σα ενδιαφέρει η δράση μα και θα δείτε περισσότερε πληροφορίε για τα προγράμματά μα. Είναι ήδη συμπεράσματο. Θέλω να τονίσω ότι από τη δική μα την οπτική γωνία βλέπουμε να υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ε, αναχαιτήσουμε τι τάσει προστατευτισμού και να προωθήσουμε ω κινητήριο δύναμη το εμπόριο για την βιώσιμη ανάπτυξη και να στραφούμε στην οικονομική ανάπτυξη και την ευμάρεια. Θέλουμε να συνεχίσουμε τι συζητήσει μαζί σα και πέραν αυτή τη ακρόαση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Πιλάλ, επικεφαλής ε, της, ε, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Πολιτικής και ε, Διαχείριση Πολιτικής. Η εμπειρογνωμοσύνη του κυρίου πιλάλ έχει να κάνει με εμπορικά ζητήματα για την ανάπτυξη, το εμπόριο και σε ό,τι αφορά κυρίως την Αφρική και τις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Έχετε το λόγο, κύριε Βιλάν. Δόκτωρ Βιλάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρευρεθώ εδώ σήμερα. Είναι σαφές νομίζω και από τη συζήτηση σήμερα το πρωί ότι το Aid for Trade αποτελεί ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, μια πάρα πολύ χρήσιμη προσέγγιση αν θέλετε. Υπό την έννοια αυτή θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δευκρινίσουμε ότι βοήθησε και την, στην εστίαση της προσοχής μας στο εμπόριο, στο αποτελεσματικό εμπόριο και στις ε, θετικέ συνέπειες που μπορεί να έχει το εμπόριο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό στην παρούσα φάση, γιατί και αυτό αναφέρθηκε ότι υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Το είπε και η κυρία Γιάγκερ σε ό,τι αφορά την εξάλληψη των ανισοτήτων. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις ανησυχίες στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που ενέχει το εμπόριο. Το εμπόριο δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Το θέμα είναι τι ωφέλη θα μπορούσε να έχει. Αν ο κόσμος δεν έχει την αίσθηση ότι το εμπόριο τον ωφέλει ή ότι μάλλον α, οξύνει τις ανισιότητες, φυσικά δεν θα το υποστηρίξει. Θα είναι μεγάλες οι ανησυχίες το Aid for Trade λοιπόν αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να γίνει πιο ομαλή αυτή η διαδικασία και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην αρχή του Aid for Trade. Αναρωτιέμαι κατά πόσο έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το εμπόριο. Γιατί όταν συζητάμε το Aid for Trade μιλάμε για την περιφερειακή ε, ενοποίηση, ανάπτυξη υποδομεών, ανάπτυξη θετικών ε, ρυθμιστικών πλαισίων. Το θέμα λοιπόν της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαδικασίας ε, βιομηχανοποίησης που περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες, ο ρόλος του ιδιωτικού κλάδου που αναφέραμε, αλλά και ο ρόλος των επενδύσεων. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Aid for Trade και αυτό, ξέρετε, ξεπερνάει κατά πολύ την στενή εμπορική ατζέντα. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα του Aid for Trade, αλλά να μην δίνεται η λανθασμένη εντύπωση ότι μιλάμε μόνο για το εμπόριο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα θέματα που μας αφορούν και ουσιαστικά το Aid for Trade το κατανοεί ο καθένας λίγο διαφορετικά και οι δωρητές και οι χώρες που λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλες οι χώρες χρειάζονται να αναπτύξουν μια στρατηγική aid for trade. Αυτό το ζητάνε, το ζητούν οι δωρητέ. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια στρατηγική ανάπτυξη. Και έτσι λοιπόν το aid for trade μπορεί να μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε στι προτεραιότητες μας, αλλά αναρωτιέμαι κατά πόσο, μήπως στην παρούσα φάση, ε, αποτελεί, αν θέλετε, και κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο και παρόλα αυτά απαιτείται. Αυτό αποτυπώνεται και στην εμπορική ατζέντα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι ακριβώ είναι το Aid for Trade σήμερα. να θυμόμαστε ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε στα μέσα της διαδικασία του 2000 με την κρίση κτλ. Οι συζητήσει όμω σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά τι επενδύσει, την ανάγκη ε, προσέλκυση άλλων μεθόδων χρηματοδότηση κτλ. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, σε ό,τι αφορά τι επιδοτήσει, σε ό,τι αφορά τον παράγοντα μόχλευση και τη χρηματοδότηση. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ουσιαστικά η βοήθεια, το aid, είναι ένα μικρό κομμάτι μόνο του aid for trade. Όταν μιλάμε λοιπόν για τη μεταρρύθμιση της δικασία του aid for trade, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το aid, η αρρωγή, είναι ένα μικρό κομμάτι και ποια μπορεί να είναι η επίδραση, ο αντίκτυπος του aid for trade. Αυτό συζητιέται και στην ε, ατζέντα για το 2020. Να πούμε λοιπόν ότι περιλαμβάνεται το θέμα της μεικτής χρηματοδότησης, αναφέρθηκε επίσης ο ρόλος ε, της ιδιωτικής χρηματοδότησης, το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα του κινδύνου και της ε, εξασφάλισης της ασφάλειας. Το θέμα της προώθησης των εξαγωγών, όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν και νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το EFSD, αλλά και το δεύτερο πυλώνα που είναι η αρρωγή ουσιαστικά που θα μπορούσε mm. να ενταχθεί στα παραδοσιακά εργαλεία του Aid for Trade, αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον στον τρίτο πυλώνα. Να σκεφτούμε λοιπόν τα θέματα χρηματοδότηση των εμπορικών ζητημάτων. Αυτό, όπω σα είπα, ξεπερνάει τα όρια του εμπορίου. Είναι πολύ πιο ευρύ θα πρέπει να κοιτάξουμε και το ποιον υποστηρίζουμε ανά πάσα στιγμή. Αναφέρθηκε αυτό από έναν συνάδελφο. Μιλάμε για υποστήριξη μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί. Μήπως ε, δεν πρέπει να υποστηρίζουμε ουσιαστικά το δικό μας ιδιωτικό κλάδο, αλλά εκ παραλλήλου. Η πρόθεση και του ευρωπαϊκού ιδιωτικού κλάδου έχει ε, σχετίζεται με τι 45 ε, ε, επενδύσει, Αυτή η διασύνδεση δηλαδή με τι αναπτυσσόμενε χώρε θα έχει αρκετικά αυθεντικό αντίκτυπο και με τι ε, αναπτυσσόμενες χώρε. Υπάρχει λοιπόν προφανώ ένα προφανέ συμφέρον για την υποστήριξη του ιδιωτικού κλάδου, όχι μόνο στι αναπτυσσόμενες χώρε αλλά και στι δικέ μα χώρε. Υπάρχουν μεγάλα ωφέλη. Αποφεύγοντα φυσικά τι επιδοτήσει και τη κρατική ενίσχυση προς τις ε, δικές μας επιχειρήσεις και την ε, μετατροπή του Aid for Trade σε ένα εργαλείο αποκλειστικά για την υποστήριξη των δικών μας επιχειρήσεων, γιατί αυτό φυσικά στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Άρα, υπό πληθιά ευρεία έννοια, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ανακατασκευάσουμε την ιδέα του Aid for Trade, να κλείσω με το στοιχείο της βιωσιμότητας της αηφορίας, το οποίο ενδεχομένω να μην έχει τονιστεί επαρκώς στη συζήτηση για το Aid for Trade. Το έχουμε ακούσει κάπως από γερμανική άποψη. αλλά στην αναθεωρημένη στρατηγική για το Aid for Trade θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο πώς προωθούμε το βιώσιμο εμπόριο. Για να υπάρχουν βιώσιμες εμπορικές πρακτικές, θεμητές εμπορικές πρακτικές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και τέλος, έχουμε και το θέμα των φίλων. Πριν το καλοκαίρι έγινε μια πολύ σημαντική διάσκεψη εδώ στις Βρυξέλλες με το ITSA και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το ρόλο των γυναικών στο εμπόριο. Νομίζω ότι η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει να ενταχθεί πολύ πιο ευρέως ε, στην Aid for Trade, όπως και το θέμα της Ενδίας ήταν στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τις τρεις μοναλίστες για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Κυρία Γιάκερ έχει ε, σκοπό να αποχωρήσει σε μερικά λεπτά, οπότε αν έχετε κάποιο, κάποια ερώτηση που απευθύνεται στην ίδια, ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί. Για να δω λοιπόν, η κυρία Χάουταλα νομίζω θα ξεκινήσει Έχω για την κυρία Γιάγκερ μία ερώτηση ε, σας άκουσα, ευχαριστώ πολύ, πολύ προσεκτικά όπως όλοι, γιατί παρουσιάσατε τα νέα στοιχεία στην αναθεωρημένη στρατηγική για το Aid for Trade και πρέπει να σας πω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία ανακοίνωση έτσι ώστε να περάσει το μήνυμα και να συζητηθεί και από το κοινό και από τους θεσμούς και από τα ε, αρμόδια όργανα. Πώς μπορείτε να το πείσετε, να πείσετε λοιπόν τον κύριο Τίμερμανς να γίνει ανακοίνωση και όχι κάποιο ε, έγγραφο ενδοϊπηρσιακό. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ερώτηση. Άκουσα τις παρουσιάσεις και θα ήθελα να μου πείτε ποια βλέπετε εσείς να είναι η ισορροπία μεταξύ της δικής μας στρατηγικής για το Aid for Trade και τις εθνικές στρατηγικές για τις ε, εμπορικές δράσεις και τις αναπτυξιακές δράσεις που συνήθως προωθούν τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας. Και μια τρίτη ερώτηση προς την Κομισιόν, κυρία Κύρτονταλ. Ναι, για τη νέα στρατηγική Είπατε πως έχει γίνει μια απογραφή και η αξιοπρεπής εργασία είναι από αυτά που θέλετε να επιτύχετε. Δηλαδή να αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά ε, προωθώντας τα δικαιώματα. Επίσης, οικοδόμηση δυναμικού των εμπλεκομένων και ξέρουμε ότι εκεί βρίσκεται η αδυναμία πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, το οποίο δεν επιτρέπει ουσιαστικά αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και θέσεις εργασίας. Έχετε λοιπόν κάποια συγκεκριμένη πολιτική στο μυαλό σας, ε, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος, να γίνεται ε, μεγαλύτερη συζήτηση, η οποία δεν θα παραμένει στα θέματα ρητορικής σε επίπεδο τουρκικής χώρες αυτές, αλλά πραγματικά θα ενισχύσει τις θέσεις εργασίας. Κυρία Γιάγκερ, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές πρώτα και μετά θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Οι επιτροπές σας πραγματικά στέλνουν τις πιο καλές ερωτήσεις και ελπίζω όντως πως μετά από πολλές συζητήσεις με τις σχετικές υπηρεσίες θα καταφέρουμε να λάβουμε μια θετική απάντηση και θα εκδώσουμε ανακοίνωση. Δεν έχω τελική απάντηση, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε σε όλα τα επίπεδα στη δική μας υπηρεσία πως αυτά θα πρέπει να ανακοινωθούν με έναν ισχυρό τίτλο και που θα ευθυγραμμίζονται με την ανακοίνωση για το ψηφιακό χάσμα από πέρσι και πως το Νοέμβριο ελπίζουμε πως θα το καταφέρουμε έτσι ώστε να ε, συμπίπτει αυτό χρονικά και με την, ε, τον εορτασμό της, της επαιτίου από την αρχική παρουσίαση της στρατηγικής Aid for Trade. Μαρέτα, να μας βοηθήσετε κι εσείς να πείσουμε και τους υπόλοιπους. Πάντως η προσπάθεια συνεχίζεται και κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας πληροφορήσει και θα σας ενημερώσει και γι' αυτό, αν μου δίνετε την άδεια. Και δεύτερον, ναι, ναι, πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο με τα κράτη-μέλη. Ξέρετε πως έχουμε μια μοναδική δυνατότητα τώρα στα πλαίσια της συνένεσης και στα πλαίσια της εφαρμογής του θεματολογίου του 2030 μπορούμε να το πετύχουμε. Επίσης, κοινό προγραμματισμός. Εκεί πραγματικά έχουμε ε, μεγάλο πεδίο να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Και το blending επίσης θα πρέπει να κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε για να εναρμονίσουμε αυτά τα στοιχεία και αποκοινούμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε έτσι ώστε ελπίζω να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις δράσεις μας και να πολλαπλασιαστεί η θετική αποτελεσματικότητα αυτών. Οπότε όταν μιλάτε με τους συναδέλφους σας παρακαλώ να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό. Και για την αξιοπρεπή εργασία είναι κάτι το οποίο προωθώ εδώ και χρόνια. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τη διαβούλευση, να δούμε σε ποιο κεφάλαιο θα το εντάξουμε είναι στις εξειδικευμένες ε, προγραμμα... Ε, δηλώσεις προγράμματος, είναι ε, σε κάποιο άλλο κομμάτι στην ανάπτυξη δυναμικού, δεν ξέρω, είναι ακόμα νωρίς, πάντως σίγουρα θα μπει στην όλη διαδικασία και θα κάνω ό,τι μπορώ από την πλευρά της Γενικής Διεθνής ΔΕΒΚΟ έτσι ώστε αυτό να έχει το ρόλο που του αξίζει στη νέα στρατηγική. Ως εργαλείο όμως προγραμματισμού δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ακριβώς πώς θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γιάγκερ. Να περάσουμε λοιπόν στον αρχικό κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Αρένα θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έκανα την ερώτηση στην κυρία Γέγκερ γιατί πιστεύω πως είναι μια πιο πολιτική ερώτηση. Έτσι θα τη θέσω. Θα ήθελα να πείτε γιατί η στρατηγική ονομάζεται Aid for Trade και δεν ε, ονομάζεται, όπως είπε κάποιος στο πάνελ, στρατηγική με τίτλο «Το εμπόριο, εμπορική πολιτική που έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση». Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Η στρατηγική λέγεται Aid for Trade. Υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας και πρέπει να το τονίσουμε. Πρέπει να επανατοποθετήσουμε την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη πώς μπορούμε να την πετύχουμε μέσω εμπορικής πολιτικής. Για τις αφρικανικές χώρες σήμερα υπάρχει το εξή ερώτημα. Η προτεραιότητα κάποιων χωρών σε παραγωγικό επίπεδο ποιο είναι να συμμορφωθούν με, τα, ε, φυτο, τις φυτογειονομικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτυχθούν περισσότερο ή θα πρέπει περισσότερο να εξετάσουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που κάνουν σε εσωτερικό και περιφερειακό επίπεδο μέσα στην Αφρική για να βελτιώσουν τις συναλλαγές με τα γειτονικά τους ε, χώρα. Για παράδειγμα, ε, η Δυτική Αφρική, η περιοχή της Νότιου Αφρική, Νότιου Αφρικής, Ανατολικής Αφρικής. Δηλαδή, το Aid for Trade. Ποια είναι η προτεραιότητα? Να στηρίξουμε project στις χώρες αυτές για να εξάγουν προς την Ευρώπη. Δηλαδή, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους δικούς μας υγειονομικούς και φυτογειονομικούς κανόνες γιατί είναι το πρώτο εμπόδιο για να εξάγει κανείς στην Ευρώπη. Η απόσταση μεταξύ αυτών των χωρών και των τρόπων που παράγουν και των απαιτήσεων που έχουν οι Ευρωπαίοι σε φυτογειονομικό επίπεδο είναι τέτοια που χάνουν χάνουν την περιφερειακή ανάπτυξη για να πετύχουν εξαγωγές προς εμάς. Αυτό είναι η αναπτυξιακή ε, προκλητική. Αν αντίθετα η στρατηγική ήταν κάπω διαφορετική. Μία εμπορική πολιτική υπέρ τη ανάπτυξης θα είχαμε λάβει τελείω διαφορετικέ κατευθύνσεις με εμπορικές συμφωνίες με την Αφρική πολύ διαφορετικέ από αυτές τι οποίες υπογράφουμε σήμερα που είναι σήμερα διμερεί μεταξύ κρατών μελών εννοώ δηλαδή κρατών μελών με αφρικανικά κράτη που καταστρέφουν την περιφερειακή ανάπτυξη και εδώ έχω μια πρώτη δυσκολία με το Aid for Trade και θα ήθελα να την επαναπροσδιορίσουμε όπως είπατε και εσείς κύριε εμπόριο προς όφελος ανάπτυξης. Δηλαδή είναι μια τελείως διαφορετική νοτροπία για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Επίσης, λέγοντας Aid for Trade, αυτή τη στιγμή τονίζουμε την πτυχή Aid, βοήθεια. Δηλαδή, λέμε είναι αποτελεσματική η αναπτυξική βοήθεια όταν μιλάμε για εμπόριο. Ή χρειαζόμαστε παραπάνω πόρου για το κομμάτι που είναι βοήθεια, aid, και λέμε με του επιπλέον πόρους θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα και ίσως να κατευθύνουμε προς το εμπόριο, αλλά μην ξεχνώντα την υγεία, την παιδεία, τα πρωταρχικά στάδια τη ανάπτυξης, γιατί σήμερα βλέπουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία λέει θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια Πρώτον, για να μην έχουμε μετανάστευση. Οπότε, σύνορα για να μην φτάνουν οι ξένοι στην Ευρώπη. Και δεύτερον, βοήθεια έτσι ώστε να μπορούν να εμπορεύονται με την Ευρώπη. Για μένα αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Ή θα πρέπει να πούμε προπολογισμοί αναπτυξιακοί και τους στέλνουμε και τους ενισχύουμε ή πάβουμε να θέτουμε το στόχο μόνο στο πόσο αποτελεσματική θα είναι η βοήθεια αυτή. Επίσης, θεμελιώδη δικαιώματα. Πώς μπορούμε στο πλαίσιο αυτή τη στρατηγική, Aid for Trade να αντιμετωπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές και με ποιο τρόπο θέτουμε τους ε, επενδυτές ενώπιον των ευθυνητών. Πρόσφατα είχα πάει στο Μαρόκο σε αποστολή και οι Ευρωπαίοι πρέσβοι στο Μαρόκο μας είπαν να συναντήσετε επιχειρήσεις για να δείτε πώς θα αναπτυχθεί η χώρα. Πολύ ενδιαφέρον. Και τι συναντήσαμε, Γάλλους στο Μαρόκο. Λες και δεν υπήρχαν Μαροκινοί στο Μαρόκο. Μα ήταν περίεργο. Εκτός μικροφώνου. Νομίζω πως το σημείο αυτό θα το αφήσουμε. Είναι πολύ περίεργο. Εμείς ξεκινάμε από την αρχή πως η ανάπτυξη στις χώρες αυτές θα γίνει από εμά και όχι από τους ίδιους. Οπότε τι ζητάμε από τους δικούς μας επενδυτές, γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το σχήμα, το οποίο δεν είναι το δικό μου, αλλά τι τους ζητάμε, όχι να κάνουν απλώς business, αλλά να φέρουν την ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι το οποίο θα επιβάλλουμε μέσω των δικών μας εμπορικών συμφωνιών. Ανοιχτό το θέμα λοιπόν, αλλά θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απάντησή σας και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τόσο είπε ο πάνελιστ από τη Γερμανία σχετικά. And, ε, Σας ευχαριστούμε κυρία Χόιμπρουφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Μαρία Αρένα και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πάντα θεωρούμε ότι το εμπόριο ουσιαστικά γίνεται σε διεθνές επίπεδο εδώ με την Ευρώπη. Αλλά εγώ κοιτάω και το περιφερειακό εμπόριο, το κατά πόσον ε, οι περιφέρειες είναι πιο μικρές περιφερειές ή πιο μεγάλες όπως και εδώ για παράδειγμα Ανατολική, ε, Δυτική, Βόρεια, Νότια Αφρική. Κατά πόσον ε, υπάρχει αυτή η διάθεση να διαμορφώθει σε τέτοιο επίπεδο το εμπόριο. Η κυρία Γιάνκερ είπε ότι υπάρχουν χώρες, για παράδειγμα, όπου η απελευθέρωση του εμπορίου ε, ουσιαστικά βοήθησε τον κόσμο να ξεπεράσει ε, την ένδια. Ε, θα με ενδιαφέρει να ακούσω παραδείγματα. Για παράδειγμα στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ προστατευτική η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το εμπόριο μέχρι ότου ξεκίνησε τη δική της ε, παραγωγή, μέχρι ότου πραγματικά ήταν ανταγωνιστική στο παγκόσμιο εμπόριο. Τότε ξεκίνησαν να ανοίγουν τις αγορές τους. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η απελευθέρωση είχε λάβει χώρα προηγουμένως η σε ό,τι αφορά τις εμπορικές ε, ε, συμφωνίες. Όταν ε, ασκούμε εμπόριο εκεί, ουσιαστικά μας ενδιαφέρουν οι πρώτες ύλες, αλλά τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να υποστηρίξουμε τις παραγωγή στις χώρες αυτές, όταν δεν προστατεύουμε καθόλου την παραγωγή. Είναι λοιπόν υπάρχει μια αντίφαση. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε εκεί τη μεταποίηση στις χώρες αυτές. Πραγματικά λοιπόν αναρωτιέμαι το τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δόκτωρα Μπιλάλα, πολλά προβλήματα αναφέρατε στην παρέμβασή σας για το γεγονός. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε ότι υπάρχει απομόνωση πολυκόσμου. κόσμου. Ίσως λοιπόν το εμπορικό ισοζύγιο να στέκει σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Πολλά προβλήματα αναφέρεται και θα ήθελα να τονίσω ένα εξ αυτών σε ό,τι αφορά το στοιχείο της βιωσιμότητας, το οποίο και τονίσατε. Το οποίο δεν τη χάνει σωστή διαπραγμάτευση, δεν τη χάνει τη αρμόδια προσοχή. Αλλά και όπω είπε η κυρία Αρένα, και εσεί μιλήσατε για την εταιρική ευθύνη. Πώ θέλουμε να πετύχουμε πιο πολύ εταιρική ευθύνη. Αν το θέμα τη κοινωνική ευθύνη το αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων για το περιβάλλον, για το κλίμα, για τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Αν το αφήσουμε σε εθελοντικό επίπεδο, τα πράγματα θα είναι λίγο ρευστά. Θα αναλυφθεί καν αυτή η ευθύνη. Πώ θα βρούμε λοιπόν δεσμευτικού ε, κανόνες. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να ακούσω απαντήσει. Charles please. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθυστέρησα. Οπότε ίσως αυτά που θα θίξω να αναφέρθηκα κανένα έλλειπα Εάν συμβαίνει αυτό, να μου το πείτε. Έχω ερώτηση για τις βάσεις επί των οποίων ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΑΚΕΑ στην Αφρική. Οι διαπραγματεύσεις αυτές βασίζονται στο άρθρο 24 του ΓΚΑΤ, της Συμφωνίας ΓΚΑΤ. Σε μια εποχή όμως που το εμπόριο ήταν διοργανωμένο σε διεθνέ επίπεδο μεταξύ χωρών που είχαν περίπου παρόμοια παραγωγή. Σήμερα τον να έχουμε διαπραγματεύσει μεταξύ εμπορικών εταίρων που έχουν αποστάσει στην παραγωγή τους αξιοσημείωτες οδηγεί στην ερώτηση εάν μπορούμε να βασιζόμαστε ακόμη στο άρθρο 24 στι διαπραγματεύσει αυτές. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη ερώτηση και κατά τα άλλα μου δημιουργεί κάποια δυσαρέσκεια το ότι το άρθρο 24 χρησιμοποιήθηκε στην αρχή των δημοκρατήσεων όταν υπήρχε μια μη παραδεδεγμένη ε, διαφωνία μεταξύ του Λουί Μισελ και μία ε, ε, άποψη φιλελεύθερη ε, και περιορισμένη. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τις αφρικανικές χώρες να ανοίξουν τις, υπερο... τις αγορές τους. Η δυσαρέσκειά μου λοιπόν ξεκινάει από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις θεωρώντας ότι είχε γίνει σωστά ο σχεδιασμός του αρχικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν μπορεί να ανατρέψει τις διεθνείς συμφωνίες που ήδη προβλέπονται, όμως θα μπορούσε να προωθήσει πλέον εμπορικές συμφωνίες στη βάση του εμπορίου που να είναι τουλάχιστον ε, βασισμένες στην ισοτιμία. Ως φιλελεύθερο είμαι υπέρ της προθεση του εμπορίου, αλλά δεν πρέπει λίγο να γίνει ο απολογισμός των προστατευτικών μέτρων που έχει λάβει η Ευρώπη από τότε που άρχισε να υπάρχει και το τι είναι διδεθειμένη να παραχωρήσει στις χώρες με τις οποίες διαπραγματεύεται. Ιδίω για τι συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση. Είναι θέμα δικαιοσύνη αυτό και θα έπρεπε να μπει στην όλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κανένας άλλος βουλευτής θα ήθελε να πάρει το λόγο. Το ερώτημα του κυρίου Γκέρενς ενδεχομένω να απευθύνεται κυρίως στο πρώτο πάνελ, ΠΟΕ και ΟΣΑ. Αν θέλετε να απαντήσετε. Μπορείτε να πάρετε το λόγο πρωτού κάνουν καταλητικά σχόλια οι πανελίστες του δεύτερου πάνελ. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, με πιάσατε. Απροετοίμαστο. Νομίζω ότι για κάποια από τα ζητήματα που αναφέρατε, ένα από αυτά ήταν πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε μόνο το εμπόριο σε ό,τι αφορά τη διάσταση του Νότου και του Βορρά, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική και άλλε περιφέρειε. Το εμπόριο έχει να κάνει πιο πολύ με την ανάπτυξη. ανάπτυξη η εμπορική ανάπτυξη είναι στο Νότο, Νότος-Νότος. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τις στρατηγικέ τις οποίες έχει υπόψη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φυσικά αυτό παίρνουμε ω σημείο αναφορά. Η ικανότητα, το δυναμικό το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε. Να δούμε ποιες είναι το δυναμικό λοιπόν για το εμπόριο σε συνολικό επίπεδο. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά κάποια περιφέρεια μόνο. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 24. Να πω δύο λόγια. Θα συνεχιστούν ε, οι συζητήσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ. Μία από τις συζητήσεις που γίνονται είναι για την διατάξεις ειδικής προνομιακής μεταχείρισης. Εδώ υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και προοπτικές μεταξύ των μελών του ΠΟΕ. Κάποια από τα σχόλια που ακούσαμε ισχύουν, αλλά άλλοι αντιθέτως τα διατείνονταν ότι ο τρόπος ανάπτυξης του δυναμικού θα ήταν ακριβώς η απελευθέρωση, η ανάληψη των δεσμεύσεων στα πλαίσια της συμφωνίας για την ευκόνιση του εμπορίου, για την ανάπτυξη εμπορικού δυναμικού δυνατότητα εξαγωγής. Δυνατότητα εξαγωγής έχει να κάνει βασικά με τη δυνατότητα εισαγωγής, γιατί αν μπορεί κανείς να εισάγει ε, σωστά, θα μπορεί να παράγει σωστά και να εξαγάγει αποτελεσματικά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές και διαφορετικές απόψεις, οι οποίες αποτυπώνονται και εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και στον ΠΟΕ. Ναι, θα πρέπει προφανώς να συνεχίσουμε τις συζητήσεις στα πλαίσια της Επιτροπής. Τώρα οι πανελίστες, αν θα θέλουν να πάρουν το λόγο για να απαντήσουν τρεις, ε, τρία λεπτά ο καθένας. Να ξεκινήσει ο κύριος Λέφλερ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Κυρία Αρένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Δεν θα τη σχολιάσω από πολιτική άποψη, γιατί αυτό δεν είναι το καθήκον μου, δεν είναι ο ρόλος μου. Αλλά να σας πω ότι προφανώς από γερμανική προοπτική μετά από 15 χρόνια ασθενή συνεργασίας με τον ιδιωτικό κλάδο. Σε ό,τι αφορά εμπορικά ζητήματα, αυτό που διδαχτήκαμε είναι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε. Προσαρμοστήκαμε λοιπόν και έτσι έχει καταρτιστεί μια νέα στρατηγική η οποία έχει έντονο προσανατολισμό στην ανάπτυξη. Και πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, ικανότητες, τις δυνατότητες, το δυναμικό των δομών μας στις τρίτες χώρες προκειμένου να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν τους δικούς τους όρους και να μπορέσουν να πετύχουν ένα συμβιβασμό ο οποίος θα είναι ωφέλιμος αμοιβαία, αμοιβαία επωφέλης ως ε, εμπειρογνώμονας για θέματα ανάπτυξη και ως οικονομολόγος Προφανώς ε. θα σας πω ότι αυτά είναι τάσεις οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ύστερα, όντως, στα πιο πολλά προγράμματα κοιτάμε και τον προσανατολισμό στο εμπόριο. Αλλά Θέλουμε να υπάρχει και ενισχυμένο εμπόριο σε κάποιες περιφερειές. Βλέπουμε λοιπόν τι περιφερειές και οι χώρες διαφέρουν. Και τίνουμε να εξετάσουμε την Αφρική ως ένα στοιχείο. Δεν ισχύει αυτό. Για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στην Ανατολή από ό,τι αλλού. Ε, ο κόσμος λειτουργεί, εργάζεται με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να το εμπιστώσουμε αυτό. Αναφέρεται λοιπόν πράγματα στα οποία πιστεύουμε και τα οποία κάνουμε. Αλλά φυσικά υπάρχει και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι ευρωπαϊκές πολιτικέ και πάλι έχετε και εσεί τα δικά σα καθήκοντα και το δικό σα ρόλο. Μπορούμε πάντα λοιπόν να αναλογιστούμε και να αναλογιζόμαστε και να εξετάζουμε πώ έχει κατάσταση και πώ μπορούμε να δώσουμε στις ε, χώρε εταίρου δυνατότητα βελτίωση τη πολιτική τη. η Κίνα. Αυτό είναι πολύ προσωπικό βέβαια, αλλά πάντα και διαρκώ εξετάζουμε την περίπτωση τη Κίνα και προφανώ η Κίνα έχει επιδείξει σημαντική ανάπτυξη, αλλά εκείνα, Κίνα, όπως ξέρετε όλοι κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι τεράστια χώρη αγορά τη. Δεν είναι παραγωγή οποιασδήποτε άλλη χώρα. Έχει και πολύ διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και υπόβαθρο από ό,τι άλλε χώρε. Είναι διαφορετικό το σημείο κίνηση. Ο Σα ευχαριστώ πολύ πολλές και σημαντικές ερωτήσεις, αλλά ας δούμε το άρθρο 24. Τι σημαίνει αυτό για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τι έχουν οι κανόνες της ΓΑΤ. Αν είσαι αναπτυσσόμενη χώρα και θέλεις να κάνεις εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με κάποια άλλη αναπτυσσόμενη ε, χώρα, χρειάζεσαι να το κάνεις μέσω της σχετικής ρήτρα και αν θες να το κάνεις με μια πιο αναπτυσσόμενη ε, χώρα θα πρέπει να το κάνεις στα πλαίσια του άρθρου 24. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά κανείς μπορεί να αναρωτηθεί γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Δεν λέω πως είναι κακό το άρθρο 24, νομίζω πως είναι μια θετική ιδέα, αλλά υπάρχει αυτή η διαφορά. Τώρα, Νομίζω ότι από τι ερωτήσει σας φαίνεται πως και το εμπόριο και η αναπτυξιακή βοήθεια για το εμπόριο δεν είναι μόνο τεχνικά θέματα αλλά και πολιτικά. Αποτελούν απόρρια επιλογών. Και ξέρω από το παρελθόν κάποια παραδείγματα και ξέρω και από την Ευρώπη πως είναι ο δωρητής ο οποίος στοχεύει σε κάποια εμπορικά θέματα, τα οποία δεν είναι πάντα προς όφελος και συμφέρον της ε, χώρας που λαμβάνει την αναπτυξιακή βοήθεια. Ξέρω ότι αυτό γίνεται καμιά φορά στις ε, διαπραγματεύσεις με την Αφρική, όπου ήθελε μεγάλο θεματολόγιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, συνθήκες εμπορικής συμφωνίας, ε, εταιρικής και το θέλανε για τις κρατικές συμβάσεις και για κάποια άλλα θέματα και υπηρεσίες, όπου οι χώρες εταίροι δεν ήθελαν να κάνουν διαπραγμάτευση. Όμως κανείς δεν υποχρεώνεται, δεν έχω τα νούμερα εδώ, αλλά για τη στήριξη Aid for Trade που προσφέρεται είναι τόσο διαφορετικά τα ποσά και τα θέματα που δεν θα έπρεπε να θεωρούμε πως προσφέρεται μόνο με πολιτικό τρόπο ή στρατηγικό τρόπο δεν έχει να κάνει μόνο με την απελευθέρωση του εμπορίου και όχι μόνο με το ελεύθερο εμπόριο. Έχουμε αρκετή βοήθεια που έχει να κάνει με το παραγωγικό δυναμικό, με τις υποδομές, με το ρυθμιστικό περιβάλλον και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο απελευθέρωση και απόλυτο άνοιγμα στο εμπόριο. Είναι διαπραγματεύσεις οι οποίες στηρίζουν τις χώρες έτσι ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις δυνατότητες και τα συμφέροντος. Οπότε το Aid for Trade δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να ανοίξουμε εμπορικά κάποιες χώρες. Αυτό είναι παραπλανητικό. Και δεν νομίζω πως υπάρχει η υποχρέωση να κάνουμε μια επιλογή μεταξύ ε, βοήθειας έτσι ώστε να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να τις βοηθήσουμε για περιφερειακό εμπόριο. Όχι. Εγώ δουλεύω στην Αφρική και όλες ε, οι χώρες εκεί κάνουν και τι δύο επιλογέ. Συνδυάζουν εξαγωγέ προς την Ευρώπη και διαπεριφερειακό εμπόριο. Και θα δείτε και στο Aid for Trade ότι υπάρχουν στοιχεία που βοηθούν τις αφρικανικές χώρες να συμμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι χώρε αναπτυσσόμενε δεν είναι υποχρεωμένε να ανοίξουν τι αγορέ στι ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά αν θέλουν να στείλουν εδώ προϊόντα, βεβαίω και θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα πρότυπά μα. Το τελευταίο σημείο έχει να κάνει με τις ανησυχίε για το εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση. Δεν οδηγεί οπωσδήποτε το εμπόριο ε, στον αποκλεισμό. Όχι το εμπόριο βεβαίως δημιουργεί κατηγορίες που κερδίζουν και κατηγορίες που χάνουν. Και εδώ πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό εξισορρόπησης και το Aid for Trade μπορεί να αποτελέσει ένα μηχανισμό αλλά όχι αν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με ένα πολύ περιορισμένο ορισμό του τι αποτελεί εμπόριο. Θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί. Αυτό ήταν το βασικό μου μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρα Μπιλάλ, τώρα νομίζω πως πως μπορώ να δώσω πάλι το λόγο στον συμπρόεδρο κύριο Βίγκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ ε, ευχαριστώ πολύ όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή γιατί πρέπει να συζητήσουμε ένα κόσμο που συνέχεια μεταλλάσσεται, το εμπόριο γίνεται ψηφιακό, ο κόσμος γίνεται ψηφιακός και όλα αλλάζουν γύρω μας και εμείς θα πρέπει θα πρέπει τις παλιές έννοιες να τις γεμίσουμε με νέο περιεχόμενο. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα είναι πολύ προσεκτική, να έχει πολλά σκέλη αυτού του νέου κόσμου. Το Edge for Trade είναι κρίσιμο για την αναπτυξιακή βοήθεια και την ανάπτυξη, αλλά όχι οποιαδήποτε ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη. Θέσει εργασία και η ανάπτυξη θα τι προσφέρει. Στην Αφρική, στην Ασία, παντού, σε όλε τι αναπτυσσόμενε χώρε. Όχι μόνο κάποιες θέσεις απασχόλησης, εκατομμύρια θέσεις. Και το Aid for Trade μπορεί να αποτελέσει και ένα εργαλείο που εμέσως με τις ε, σχετικές στρατηγικές να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και σας ευχαριστώ που κάνατε τη συζήτηση ε, μεταξύ Επιτροπών Ανάπτυξης και Διεθνούς Εμπορίου.